So, ich bitte alle Kolleginnen Καλημέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να καθίσετε στις θέσεις σας, ώστε να ξεκινήσουμε. Έχουμε τώρα τη συζήτηση για το σύστημα εμπορίας εκπομπών Stop the Clock 2 ή όπως το λέμε στο κοινοβούλιο The Never Ending Story η ατέρμονη ιστορία. Καλωσορίζω τον μόνιμο εισηγητή μας. Τον και τον οικουμενικό θα έλεγα εισηγητή, καθώς τον έχουν ε, προτείνει όλες οι ομάδες ε, να αναλάβει το θέμα αυτό. Πράγμα το οποίο δείχνει βεβαίως ε, την εμπιστοσύνη της οποίας χαίρει. Κύριε Λύση, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Οι τροπολογίες που έχουν κατευθεί και που έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Καθιστούν σαφές ότι έχουμε ένα πολιτικό πρόβλημα και θα ήθελα να επισημώ ότι κάποιοι οι οποίοι ε, περιγράφουν σενάρια τρόμου ως προοπτική, καλό θα ήταν να ξανακοιτάξουν ποια είναι η πραγματικότητα. Διότι βλέπουμε μια πολύ περιορισμένη επιβάρυνση για, τις, ε, για το μεταφορικό κλάδο και τους επιβάτες. Η Ryanair, παραδείγματι, έχει κόστος 0,03 ευρώ, δηλαδή 3 λεπτά του ευρώ. Άλλες εταιρείες, λιγότερο αποτελεσματικές, μπορεί να έχουν υψηλότερο κόστος. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι κοστίζει μία ε, μακράς αποστάσεως πτήση σε μια αεροπορική εταιρεία περισσότερο από, ε, από τα 2 ευρώ. Η γερμανική, η βρετανική και ε, γαλλική κυβέρνηση ζητούν από τους πολίτες τους την καταβολή τελών όταν ταξιδεύουν από τη Φραγκφούρτη, το Λονδίνο ή το Παρίσι, πολλαπλάσιων των ποσών αυτών. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι εμπλέκονται και τρίτα κράτη. Άρα έχουμε μια πολύ ε, παράδοξη κατάσταση και θα πρέπει να φροντίσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να μην χάσουμε τον μπούσουλα, διότι δεν μπορεί εθνικά μέτρα να παρεμποδίζουν την ανάπτυξη μιας κοινή πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από τροπολογίες, 90 συνολικά για την ε, πρόταση εκθέσεως, οι οποίες καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των συζητήσεων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ακραία θέση θα έλεγα είναι αυτή του Μπασάικχουτ η οποία όμως επιμερίζει την επιβάρυνση στους διάφορους εμπλεκόμενους, όχι μόνο τις μη οργανώσεις, αλλά... Μάλλον υποστηρίζει υποστηρίζεται όχι μόνο από μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και από τις πολύ χαμηλές, χαμηλού κόστους εταιρείες, την ΕΛΦΑ, που εκπροσωπεί μεγάλο ποσοστό αυτών των αεροπορικών εταιριών. Προσπαθεί να επαναφέρει το αρχικό σύστημα η πρόταση αυτή, δηλαδή οποιοδήποτε αεροσκάφος προσγειώνεται ή απογειώνεται από ευρωπαϊκό αεροδρόμιο θα πρέπει να εφαρμόσει, να επάγεται στο αρχικό ETS, το σύστημα ανταλλαγών, όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί. Οι κυρίες Κόρχολα Γκροστέτ, ε, ο κύριος Κράμαρ και άλλοι έχουν υποστηρίξει ε, την ε, πρόταση να παραταθεί το σύστημα, η, η αρχή του stop the clock, η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα μέχρι την επόμενη συνέλευση της ΙΚΑΟ και αυτό άλλωστε υιοθέτησε και η Επιτροπή των Μεταφορών την Τρίτη. Τώρα πρέπει να τα συστήσουμε όλα αυτά. Γιατί έχουμε λίγο πολύ να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Από τη μία στην άλλη θέση το να βρούμε συμβασμούς θα είναι ισοδύναμο το να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βρει λύσεις όχι full scope, ούτε stop the clock, αλλά airspace. Έχουμε αντιμετωπίσει αντιστάσεις βεβαίως, έχουν εκφραστεί αντιστάσεις, ιδιαίτερα οι αεροναυπηγικές εταιρείες όπως η Airbus έχουν αντιδράσει πάρα πολύ και άλλοι βεβαίως μας έχει πει ο πρόεδρος ότι απέστειλε επιστολή στους Κινέζους, στην κυβερνητική κυβέρνηση Airbus, όπου δείχνει πως θα έχουμε σοβαρή αντιπαράθεση. Αν λοιπόν ξεκινάμε έτσι και αν πρέπει να πείσουμε την Κίνα ποιο είναι το δικό μας συμφέρον και να το ακολουθήσει η, Ευρω... η Κίνα, τότε ασφαλώς θα είναι δύσκολος ο αγώνας. Ο Ντέιβιτ Κάμερον στις συνομιλίες του με την Κίνα τοποθετήθηκε με πολύ έντονους όρους ως προς την κατάσταση αυτή για την ε, Airbus. Ε, επικαλέστηκε ακόμα και τον ε, Δαλάη Λάμα. Ασφαλώς η κατάσταση θα είναι δύσκολη. Εάν αρχίσουν οι Κινέζοι να ανατρέπουν συμβάσεις, τότε ασφαλώς θα πρέπει να τους, να τους τίνουμε και ευηγονούς από ό,τι φαίνεται. Καλύτερα να μην φτάσουμε μέχρι εκεί λοιπόν. Και γι' αυτό πιστεύω και ζητώ και την κατανόησή σας ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Εγώ είμαι ε, ως εισηγητής εκ μέρους του Κοινοβουλίου υποχρεωμένος να λάβω υπόψη τα όσα φρονούν η μεν και η δε, συναδελφοί μέσα στο Κοινοβούλιο. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα βέβαια με, την, ε, με τον όγκο των τροπολογιών να φτάσουμε ε, στην Ολομέλεια εγκαίρως με την αρχική πρόταση εκ δηλαδή. Θα έχουμε πολύ περιορισμένο ε, χρόνο, δεν θα φτάσουμε δηλαδή στην Ολομέλεια πριν από τις ευρωεκλογέ. και άρα και ιδιαίτερος καθώς πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη θέση της Επιτροπής των Μεταφορών αλλά και της Επιτροπής ε, ε, Βιομηχανίας η οποία όμως ακόμη δεν έχει λάβει απόφαση αυτή την ώρα μάλλον τη λαμβάνει και δεν είμαι ενήμερο για το τι θα κάνει. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν και αυτές τις τοποθετήσεις. Θα κάνουμε συνεδρίες των σκιωδών εισηγητών σήμερα το απόγευμα. Θα δω τι είδου δυνατότητες για συμβασμού υπάρχουν, ώστε, και δεσμεύομαι εγώ ω εισηγητής, να προχωρήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό εφόσον υπάρχει περιθώριο κινητικότητας. Θα δούμε. Εχθές συζήτησα με τους κοιόδης Έκανα μια αρχική πρόταση, ένα συλλογισμό χωρίς να μπορώ να πω ότι έγινε δεκτή ομόφωνα και χωρίς να μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από την κατάσταση που αντιμετωπίζω, δεδομένου ότι έχουμε <laughs> δημοκρατία και είμαι και εγώ δημοκράτης πρέπει να δεχθώ τις διαφορετικές απόψεις. Η Επιτροπή των Μεταφορών ιδιαίτερως με προβληματίζει, αλλά θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε στο δυνατόν περισσότερες από τις δικές τροπολογίες και, σε αυτό το πακέτο, και από αυτές τις τροπολογίες στο πακέτο. Ιδιαίτερα παραπέμπει στις θέσεις της ΙΚΑΟ και της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΤΡΑΝ, ε, ε, ζητεί την παράταση του Stop the Clock και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια θα είναι η δυνατότητα για παράταση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το 2016 όπως ζητάει η Επιτροπή των Μεταφορών. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη μιλάει για ένα χρόνο παράταση ως ε, προς τις ευρωπαϊκές πτήσεις στο, στο σύστημα ανταλλαγή των εκπομπών και εάν δεχόμαστε αυτή τη λύση της ε, ετήσιας παράτασης θα πρέπει να ξέρουμε σε τι χρησιμεύει. Εγώ θα έλεγα και θα το πω και στην ψηφοφορία όταν έρθει η ώρα ότι χρειάζεται αυτή η παράταση για να βελτιωθεί η αποδεξιμότητα αυτής της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Αέριο Χώρο, το Airspace Approach να γίνει δηλαδή πιο ε, κατανο... ευρέως κατανοητή και αποδεκτή αυτή η πρόταση. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε πάντοτε όταν ε, θέλουμε να πείσουμε για τις δικές μας θέσεις και μάλιστα όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο πρέπει να δείχνουμε περισσότερη διαλλακτικότητα. Ένα άλλο ζήτημα λοιπόν και σημείο καμπής πιστεύω θα είναι το να καταφέρουμε να πείσουμε τα κράτη, να υποχρεώσουμε καλύτερα τα, τα κράτη να διαπραγματευτούν το ζήτημα των ε, εσόδων από τις ανταλλαγές εκπομπών. Ένα ζήτημα πολύ κρίσιμο, διότι τα τρίτα κράτη λένε «Α, ναι, κάτι κάνουμε για τις ε, ε, για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά δεν ορίζεται πουθενά στην νομοθεσία το που θα αξιοποιούνται τα έσοδα αυτά. Ε, είναι κάτι όμως το οποίο το Κοινοβούλιο έχει συζητήσει από την αρχή. Νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε στο διεθνή διάλογο με τη βιομηχανία, με το βιομηχανικό κλάδο, με τους Αμερικανούς, με τη διεθνή διάσκεψη για το κλίμα, το adaptation και mitigation μπορούμε να το συζητούμε και φαντάζομαι ότι στις διεθνείς διασκέψεις, ε, εν ώψη της διασκέψης των Παρισίων συγκεκριμένα, στο Παρίσι ή ε, ε στο, καθοδόν προς το Παρίσι θα μπορούσαμε να πείσουμε τον Επιτρόπο γιατί συζητάει για τις ε, εκπομπές αλλά δεν μιλάει για το οικονομικό σκέλος. Μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη δεν είναι διατεθειμένα να συστήσουν το θέμα αυτό λοιπόν και εκεί νομίζω βρίσκεται και το κλειδί της λύσης αυτής της υπόθεσης. Ήταν αρχικά εξ αρχής η θέση του Κοινοβουλίου αυτή να ε, τεθεί το ζήτημα αυτό και έχουμε πει εξ αρχής ότι αν το Συμβούλιο δεν θέλει να, να προχωρήσει το θέμα αυτό έχει δογματικές θέσεις και εμείς θα πρέπει να κινηθούμε με περισσότερο ρεαλισμό. Έρχονται λοιπόν λένε τις θέσεις τους διάφοροι υπουργοί κάθε φορά και πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί τέλος σε αυτή την ε, κατάσταση, την ακίνηση από πλευράς του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι και σκιώδη στο θέμα αυτό και θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι τις θέσεις σου στα όσα μας είπες. Έχει περάσει αρκετό καιρό που δουλεύουμε το θέμα αυτό, από το 2008. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχουμε ξεκινήσει το ζήτημα τη επέκταση του συστήματο των εκπομπών και στι ενέργειε μεταφορέ. Έχουμε ω κοινοβούλιο εξ αρχή αναπτύξει έναν ταχύτατο ρυθμό εργασιών ε, Ήρθε η ώρα του stop the clock, όπως είπε και ο κύριος ε, Λίσε, το Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο θέτει τα προσκόμματα σε όλη την πορεία, είναι αυτό που τραβάει πίσω το τρένο θα λέγαμε και έτσι πια έχει έρθει η ώρα να προχωρήσουμε. Θα έλεγα δεν να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποιο βαθμό έχετε, τεθεί σε εφαρμογή ισχύουσα η νομοθεσία, ε, ε, τι συστήματα υλοποίηση έχουν, επιδείξει τα κράτη-μέλη, έχουν μεταφέρει το δίκαιο, έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις ή υπάρχουν κάποια τα οποία καθυστερούν ακόμη. Αυτό πρέπει να το συστήσουμε. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα κράτη συγκεκριμένα τα οποία δεν έχουν εφαρμόσει το δίκαιο ή το αγνοούν ακόμη. Γιατί ίσως είναι πολύ πιο εύκολο να, να εξασφαλίσουμε την ε, εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως λέει και ο Πίτερ έχουμε περιορισμένο χρόνο, παρά να προσπαθήσουμε να την τροποποιήσουμε. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Εξασφαλίσουμε λοιπόν την εφαρμογή της νομοθεσίας πριν προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάτι. Stop the clock υπαριθμών 1, stop the clock υπαριθμών 2. Ε, μπορεί να είναι μία λύση προσωρινή, αλλά από την άλλη δεν ξέρουμε πώς θα ξεφύγουμε από αυτή τη δύσκολη περίοδο και έχουμε και τις διεθνείς μας υποχρεώσεις εν ώψη της των Παρισίων του 2015. Είναι σαφές ότι πρέπει να αναλάβουμε και σε διεθνές επίπεδο πρωτοβουλίες. Αν όμως ε, πάμε εκεί χωρίς να έχουμε εφαρμόσει στο εσωτερικό μας την νομοθεσία που έχουμε ε, εγκρίνει, τότε δεν μπορούμε να έχουμε και επιχειρήματα για τη έσκυψη των Παρισίων. Αυτά λοιπόν, θα θέλαμε λεπτομέρειες πληροφορίες. Ποιο κράτος εφαρμόζει τι, πώς, εάν όλα τα κράτη έχουν εφαρμόσει, σε ποιο βαθμό κτλ. Και θέλουμε ονόματα των κρατών που αγνοούν την νομοθεσία. Αυτό για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ε, γρήγορη εκκίνηση ή επανεκκίνηση της ε, διαδικασίας. Κύριε uh, Ευχαριστώ. Εγώ περίμενα να ακούσω πρώτα την Φώστερ και τον Κάλαναν, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ υποστηρίζω τις προτάσεις του Λίζε, αναγνωρίζω ότι εργάζεται πάρα πολύ σκληρά για να πετύχουμε ένα συμβιβασμό σε όλο το κοινοβούλιο. Είναι δύσκολο το θέμα και υπάρχουν πιθανές επιπτώσεις αν εμείς ε, υιοθετήσουμε την πρόταση του Πίτερ και δέχομαι τις επιπτώσεις αυτές. Πρέπει να λειτουργήσουμε σαν μοχλός, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση για να πετύχουμε την συμφωνία. και δεν είμαι πεπισμένος από αυτά που λέει το ΙΚΑΟ. Αν προχωρήσουμε εμείς θα ακολουθήσουν και οι άλλοι. Ευχαριστώ. Chris. Έχουμε μια επιτροπή συνασπισμού. Ίσως θα έπρεπε να συνεννοηθείς με τις σειρέ πίσω σου για τη σειρά. Η κυρία Χάση έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σέβομαι τις εργασίες του Πέτε Λίζε και πάντα κάνει τεράστιες προσπάθειες για να διαπραγματευτεί μια καλή συμβιβαστική λύση και σε κοινοβούλιο και να υπάρξει και κοινό τόπος με το Συμβούλιο. Δυστυχώς όμως εδώ έχει, το έχει παρακάνει στην προσπάθεια του συμβιβασμού θα έλεγα. Κατά τη διάρκεια της περίοδου που είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οικονομικός γίγας και πολιτικός νάνος. Αν συνεχίσουμε εμείς να συμπεριφερόμεθα με τον ίδιο τρόπο, να νομοθετούμε δηλαδή και οι υπόλοιποι να μας πιέζουν και να διαμαρτύρονται και να μην εφαρμόζονται η νομοθετική μας ρύθμιση, τότε φοβάμαι ότι σμικρίνουμε την σημασία μας και δεν παίζουμε το ρόλο που θα έπρεπε. Δεν θα πρέπει λοιπόν εμείς να υποχωρήσουμε και να δώσουμε την εικόνα στον υπόλοιπο κόσμο ότι κάποιες άλλες χώρες διαφωνούν και αν μεγάλες επιχειρήσεις διαφωνούν με τις νομοθετικές μας ρυθμίσεις τότε τις αλλάζουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ξένες επιχειρήσεις και ξένες κυβερνήσεις λέγουν ότι είναι, ε, δεν είναι ευτυχείς με την προτινόμενη νομοθεσία μας. Εδώ και δέκα χρόνια οι πρώτες επαφές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ένας Αυστραλός πρέσβης ο οποίος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την νομοθετική μας πρόταση για τα χημικά, το REACH και η Αυστραλία ήταν εναντίον όπως και οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν εναντίον. Τι έπρεπε να κάνουμε λοιπόν. Δεν είναι η πρώτη φορά όπου διαπιστώνουμε ότι άλλες κυβερνήσεις είναι σαφώς κατά των νομοθετικών μας ρυθμίσεων. Το θέμα έχει αρχίσει λοιπόν και γίνεται συμβολικό σχετικά με το κόστος της εμπορίας ε, εκπομπών και των τελών για τις αεροπορικές επιχειρήσεις. Το θέμα όπως είπα είναι συμβολικό μιας γενικότερης κατάστασης, όχι τόσο οικονομικό. Έχω προτείνει εξ ονόματος των Πρασίνων πολλές τροπολογίες για την ενίσχυση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι καλή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτείνουν μια σαφέστατη συρρήκνωση του προγράμματος για την εμπορία των ρήπων από πλευράς της αεροπορικής βιομηχανίας στις αερομεταφορές. Αυτό ε, είναι απαράδεκτο γιατί στην ουσία δείχνει ότι υποχωρούμε άτακτα στις πιέσεις των υπολείπων χωρών. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διευρύνουμε γεωγραφικά τον τομέα ενασχόλησής μας έτσι ώστε όχι μόνο ο αδαφικός παράγων αλλά να συμπεριληφθεί και η ζώνη οικονομικής εκμετάλλευσης άνω των 200 μιλίων και τουλάχιστον το 50% των εκπομπών και από τις εισερχόμενες και από τις εξερχόμενες πτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται από το σχήμα, από το πρόγραμμά μας. Ο Πέτα Λίζε αναφέρθηκε σε κάποιες απόψεις του Κοινοβουλίου ότι τα έσοδα από τα τέλη αυτά θα πρέπει να δοθούν σε δραστηριότητες σχετικές με το κλίμα. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με αυτό. Έχω την αίσθηση ότι διεθνώς η κατάσταση θα ήταν διαφορετική αν μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έχουμε απλά με ένα νέο τρόπο να κάνουμε συλλογή τελών προς όφελος των κυβερνήσεων, αλλά ε, για την δράση για το κλίμα, για την συνδρομή στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό θα καταστήσει νομίζω καλύτερη και πιο ευνοϊκή και την στάση των ΙΠΑ και των αναπτυσσομένων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν που το Συμβούλιο δεν θέλησε να εξετάσει αυτή τη διάσταση. ένα τελευταίο σημείο. Όταν μιλάμε για συμβιβαστικές τροπολογίες θα πρέπει να ενθυμόμεθα και το Συμβούλιο ότι το Συμβούλιο δεν πρέπει να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Αν δεν υπάρξει συμφωνία ανάμεσα σε εμά και το Συμβούλιο τότε θα επανέλθει σε ισχύ η αρχική νομοθεσία. Κάλεναν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το θέμα αυτό έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον με σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις. Φυσικά από τη μία κατανοώ τη θέση του ΠΕΤΑ και των Πρασίνων που εργάζονται πάνω σε αυτό το θέμα εδώ και αρκετά χρόνια. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει επαρκώς ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ μικρό οικονομικά, το κόστος είναι λίγα ε, ε, ε, σέντ αναπτύσσει. Από την άλλη θα πρέπει να εμείνουμε για λόγους αρχής ανεξαρτήτως των συνεπειών. Οι συνέπειες εδώ είναι σοβαρές και το γνωρίζουμε. Αναφερθήκατε στην Airbus, Ξέρω ότι εμπά στο Φίλτον και στην εκλογική μου περιφέρεια απασχολεί χιλιάδες επιχειρήσεις. Και δεν θέλουμε εμείς ε, να πούμε ότι θα θέσουμε την ύπαρξή τους σε αμφισβήτηση, αλλά θα δημιουργήσουμε προβλήματα στην επιχείρηση αυτή για μικρό οικονομικό κέρδος για τα δημοσιονομικά. Αυτό θα έχει επιπτώσεις λοιπόν. Και υπάρχει και το θέμα της συμμόρφωσης. Εγώ πιστεύω στον κανόνα του δικαίου, εγώ πιστεύω στην αρχή ότι αυτή τη στιγμή γίνει δεκτή μια νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να εφαρμοστεί. Και δεν θα ήμασταν ρεαλιστές αν πιστεύαμε ότι η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα αρχίσουν να κατάσχουν ε, αεροσκάφη στη Φραγκφούρτη, στο Παρίσι, στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω ακριβώς αυτής της νομοθετικής ρύθμισης. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τις διεθνείς σχέσεις μας ε, λόγω ακριβώς αυτού του μέτρου. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές λοιπόν, άκουσα τα επιχειρήματα, ήταν λάθος που υπεψηφίστηκε η πρόταση αυτή, το είχα πει και τότε, απαιτείται ένας κάποιος συμβιβασμός να αποφύγουμε τις αρνοτικές επιπτώσεις και ελπίζω ότι οι προσπάθειες τις οποίες κάνει ο Πίτα για να υπάρξει μια συμβιβαστική λύση ε, θα αποδώσουν γνωρίζει τη στάση μας ο Πέτα, δεν θα την επαναλάβω. Απαιτείται όμως να υπάρξει μια κάποια λύση και η λύση αυτή πρέπει να βρεθεί το ταχύτερο δυνατόν, δηλαδή πριν από τον μήνα Μάρτιο. Υπάρχουν κάποιες κατευθύνσεις τις οποίες ακολουθήσουμε, θα ακολουθήσουμε, όχι εύκολες για το Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να συνεννοηθούμε και με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο. Δεν μπορώ να υποστηρίξω λοιπόν και την λεγόμενη σε εισαγωγικά προσημείωση των εσόδων. Αυτό είναι κάτι το οποίο με αφήνει αδιάφορο, δεν είμαι πεπισμένος για τα ταμεία για το κλίμα και τη μετρίαση των κλιματολογικών αλλαγών και γι' αυτό δεν θα δεχθούμε εμείς ε, την ε, ε, υποθήκευση αυτών των ποσών. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, μπας περιπτώσει περαιτέρω, αλλά όλοι γνωρίζουμε τις βασικές αρχές του καθενός μας. Ευχαριστώ. Κύριο και δεν είναι εδώ. Κύριε Φώστερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Πίτερ Λίζα. Κανένας δεν πιστεύει ότι δεν είναι δύσκολη η προσπάθεια την οποία κάνει ο Πέτα. Ένα θέμα είναι οι αρχές βέβαια, από την άλλη πρέπει να είμαστε πρακτικοί. Το θέμα εδώ είναι η επιμονή σε δογματικές αντιλήψεις όχι από πλευράς του Πετελίζε αλλά από πλευράς της Γενικής Διεύθυνσης της Κομισιόν για το Περιβάλλον που έχει γίνει τώρα Γενική Διεύθυνση Κλίματος. Ε, είναι απαράδεκτες αυτές οι θέσεις. Οι συνέπειες ε, οδηγούν σε μονομερείς ενέργειες αγνοώντας την διεθνή θέση και τις ε, αερομεταφορές. Ελπίζω στο μέλλον να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη γιατί έχουμε φτάσει με το Κοινοβούλιο τώρα σε μια πιο πολύ δύσκολη ε, ε, κατάσταση. Εγώ δεν ομιλώ εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών αλλά εξ ονόματος της ομάδας μου εκεί Νομίζω ότι η κατάσταση στην οποία έχουμε φτάσει τώρα ε, δίνει την δυνατότητα ε, να προχωρήσουμε με την ε, διάσταση stop of the clock μέχρι το 2016. Έχω καταθέσει μια τροπολογία που δεν είχε γίνει δεκτή αλλά θα σας τη διαβάσω γιατί δείχνει νομίζω το πού βρίσκονται οι προκλήσεις λόγω ακριβώς της έλλειψης μιας πραγματικής μελέτης επιπτώσεων και της δημιουργίας ε, ενός προτύπου για τη λειτουργία αυτής της διαδικασίας, η αποτυχία σεβασμού της συμφωνίας που έγινε του 2013, που απαιτεί από τις χώρες που θέλουν να εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά, να επιζητούν την αμοιβαία συμφωνία των τρίτων χωρών αναμένεται να υπάρξει βλάβη για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε εμπορικό επίπεδο ε, και στις σχέσεις με τις τρίτες χώρες, όπως επίσης και μια δημιουργία μη ανταγωνιστικού περιβάλλοντος εις βάρος των χωρών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αναβληθεί επαόριστον η εφαρμογή της συμφωνίας. Καταλαβαίνω βέβαια ότι αυτό παρουσιάζει δυσκολίες, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε τόσο ελαφρείς απέναντι στα εμπορικά μας συμφέροντα και επίσης και απέναντι στις μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις συζητούσα και στη Γερμανία που έχει τεράστιες εγκαταστάσεις η και στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο Ξέρουμε ότι έχουν υπάρξει δισεκατομμύρια δολαρίων επενδύσεων και γενικά το θέμα αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Θα πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν να κατανοήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τι έχει συμφωνηθεί στο ΙΚΑΟ, το τι συμφώνησε στο ΙΚΑΟ και το τι ήρθε και μας μετέφερε εδώ η αλλαγή ε, αυτή στη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που προσπάθησε να μας μεταφέρει με διαφορετικό τρόπο την πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο δημιούργησε δυσκολίες. Πρέπει να αναζητήσουμε μια συμβιβαστική λύση. Αν πούμε ότι θα εγκαταλείψουμε το ETS και θα συνεχίσουμε με ένα σύστημα το οποίο θα επηρεάζει αποκλειστικά τις εσωτερικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση πτήσεις, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν περιλαμβάνεται στην αρχική συμφωνία και εμποδίζουμε και τις περιφερειακές, ε, τα περιφερειακά αεροδρόμια να αποδώσουν, τις περιφερειακές επιχειρήσεις να αποδώσουν, θα επιβαρύνουμε τη λειτουργία τους ακριβώς γιατί δεν γίνεται μια λογική αξιολόγηση και το τι θα γίνει με τα πιθανά έσοδα, κοιτάξτε, αυτά είναι έσοδα από ιδιωτικές επιχειρήσεις, είναι φορολογία και θα πρέπει να δαπανώνται τα χρήματα αυτά όπως αποφασίζουν τα κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει να πηγαίνουν τα χρήματα αυτά σε οδήποτε ταμείο των Ηνωμένων Εθνών ή οπουδήποτε αλλού. Εύχομαι στον Πέτα Λίζ ε, ε, καλή τύχη και νομίζω ότι αυτή η διάσταση απόψεων ανάμεσα στους πρατίνους και τους υπολείπους πρέπει να επιληθεί. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις τις οποίες θα πρέπει να δώσουμε για να μετριάσουμε τις επιπτώσεις των εκπομπών ε, για το περιβάλλον, για τις κλιματολογικές αλλαγές, για τις εκπομπές καυσαερίων, για τις εναέριες μεταφορές, τις επίγειες μεταφορές, τις θαλάσσιες μεταφορές. Υπάρχουν πολλές προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για τη μετρίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας και όχι μόνο αυτή η οποία προτείνεται. Ευχαριστώ τον εισηγητή λοιπόν και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Κύριος Γκυμπράντη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βάσει αυτών που θέλουν ε, να παραμείνουν στο stop the clock ή να παρατείνουν αυτό το σύστημα, πρέπει να φανούμε εμείς ε, ε, πραγματιστές και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη. Το Παγκόσμιο Φόρουμ δημοσίευσε μια μελέτη σε σχέση με τις, ε, τους παγκόσμιους κινδύνους ε, για τις επόμενες δεκαετίες. Ως προς τον αντίκτυπο και τις πιθανότητες, οι κλιματικές αλλαγές είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος ε, και σε σχέση με τους υπόλοιπους μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές. Ε, λίγοι κίνδυνοι συνδέονται με την οικονομική κρίση. Ας είμαστε λοιπόν ε, σοβαροί πρώτα απ' όλα. Θα πρέπει να δείξουμε πολύ μεγαλύτερη πυγμή και ε, στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Είχαμε το σύστημα ΣΕΔΕ, ETS και είχαμε αποφασίσει να συμπεριλάβουμε και την αεροπορία. Λογικό. Πρώτα απ' όλα δεν βλέπω ούτε έναν λόγο για να αποκλείσουμε οποιοδήποτε τομέα. Δεύτερον, η πολιτική αεροπορία νομίζω είναι από τους ευκολότερους τομέας προς ενσωμάτωση, διότι ισχύουν θεμητοί όροι ανταγωνισμοί, δεν υπάρχει διαρροή άνθρακα και το καθεξής. Δεν βλέπω, ξαναλέω, ούτε ένα λόγο για να μην το κάνουμε αυτό. Δεν άκουσα κανένα ισχυρό ε, επιχείρημα ε, κατά της ε, ε, διατήρησης της προηγούμενης ε, κατάστασης, πριν το stop the clock δηλαδή. Ο κύριος Κάλλον μας μίλησε για το αντίτιμο των αρχών. Μπορώ και να το αντιστρέψω εγώ το επιχείρημά του και να του πω ποιες είναι οι αρχές ε, των τιμών που επιλέγουμε και τι μου κάνει εμένα εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση το πόσο πληρώνουμε για τον καφέ όταν παίρνουμε το αεροπλάνο ε, και ακούγοντας ε, τις κινέζικες ή τις αμερικανικές ε, αερογραμμές να μας λένε ότι επιβάλλουμε εμείς καταναγκαστικά τέλη στις στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων θα πρέπει να γίνει αποδεκτό ίσως ότι κάποια κράτη-μέλη δεν θα εφαρμόσουν αυτήν την νομοθεσία. Μα τι εστί μεγάλο νομοθέτημα, μικρό νομοθέτημα, πού ε, ε, θα τραβήξουμε τη διαχωριστική γραμμή και πού ξέρουμε ε, και πώς ορίζουμε το ότι είναι αρκετά μεγάλο για να έχει σημασία αν θα εφαρμοστεί σωστά ή όχι από όλα τα κράτη-μέλη. Το θέμα είναι ότι όταν είναι κοινοτική νομοθεσία εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη. Τελεία. Ε, νομίζω ότι το, το πιο σημαντικό αυτό είναι και εξάλλου τίθεται και βασικό ζήτημα αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δηλαδή θα χρειαστούμε τουλάχιστον ένα χρόνο για να βρούμε ρεαλιστικές λύσεις για μια, ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά αυτό πρέπει να κάνουμε και να πούμε, ε, δηλαδή τι, ότι θα εφαρμόσουμε το παλαιότερο σύστημα εάν δεν καταλήξουμε σε, σε λύση. Τι θα απειλήσετε, δηλαδή αυτό είναι το επιχειρημά σας απειλείτε ότι θα επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Ε, πρόκειται για έναν στιγνό εκβιασμό και δεν θα σταματήσει αυτό με το, την Airbus ε, αν δεν ακολουθήσουμε τη σωστή οδό τώρα, αυτή τη στιγμή. Η Βραζιλία, η Κίνα, η Αμερική ξέρουν τι κάνει η Ευρώπη, ποιο είναι το, η τεχνική της. Ε, παίρνετε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις σε κάποια μεγάλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απειλείτε ότι θα διακόψετε τις συμβάσεις μαζί τους δεν πρέπει να λειτουργούμε όπως παλαιότερα στην Ευρώπη. Θα πρέπει να συμπαραταχθούμε όλοι και να υποστηρίξουμε αυτή τη φορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω δε ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δείξει μεγάλο στένος και να μην υποκύψει σε αυτόν τον οικονομικό εκβιασμό. Ευχαριστώ. Ο Ζέπερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ότι Έχουμε να κάνουμε κυρίως με το ζήτημα εάν παίρνουμε το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση σοβαρά ή εάν υποτασσόμεθα στις πιέσεις. Όπως λένε και οι Βρετανοί συνάδελφοι, ότι πρέπει να υποχωρήσουμε. Βεβαίω μπορεί να υπάρχουν άμεσες οικονομικές επιπτώσεις, αλλά θα είναι ελάχιστη, ελάχιστο το μέγεθός τους και νομίζω ότι δεν μας προσφέρουν τίποτα αυτά που, λένε, που λέει η κυρία Φώστερ και άλλοι. Ένα λεπτό του ευρώ είναι ελάχιστο μέγεθος, μη μετρήσιμο. Και αν νομίζω η γενικότερη ζημιά είναι ένα κβαντικό άλμα σε σχέση με αυτό που μας λένε για την επιβάρυνση του οικονομικού κλάδου, τότε νομίζω ότι δεν μπορεί καν να μετρήσει στην αξιολόγηση των επιπτώσεων. Εάν όμως θέλουμε να κάνουμε αξιολόγηση των πολιτικών επιπτώσεων, τότε είναι μια άλλη ιστορία, γιατί και τα εμπλεκόμενα κράτη και βεβαίως τα ευρωπαϊκά κράτη ιδιαίτερως δεν θέλουν να προχωρήσει η Ευρώπη ενωμένη και το θέμα είναι αν μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι η Ευρώπη είναι σε θέση να προχωρήσει ενωμένη και με μια ενιαία διαπραγματευτική θέση, αν μπορεί δηλαδή να λαμβάνει αποφάσεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αποδείξουμε πρέπει να το αποδείξουμε ότι μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις, γιατί μόνο έτσι εξασφαλίζουμε και την αξιοπιστία μας στη τελευταία ανάλυση σχέση με την πολιτική για, το, για την κλιματική αλλαγή. Ιδάλλως χάνουμε κάθε αξιοπιστία και δυνατότητα να επηρεάσουμε την κατάσταση σε σχέση με τις εκπομπές στις εναέριες μεταφορές. Ο Πέτερ Λίζα έκανε πολύ καλές παρατηρήσεις, μας λέει ότι νομικά υπάρχει δυνατότητα, το έχουμε βεβαιώσει άπειρες φορές. Πρέπει απλώς να λύσουμε το πολιτικό ζήτημα. Θέλουμε να υπάρχει Ευρώπη ή δεν θέλουμε. Οι Βρετανοί φίλοι γι' αυτό έχουν επικριτική στάση, το γνωρίζουμε άλλωστε και από την ιστορία, αλλά και από τα πολιτικά τους προγράμματα, ότι η θέση τους είναι διαφορετική. Αλλά εμείς πρέπει να επιμείνουμε και να αποδείξουμε ότι το Κοινοβούλιο και αν θέλουμε βεβαίω και η Επιτροπή να, να, να υποστηρίξουμε και την πρόταση της Επιτροπής στο βαθμό που είναι ικανοποιητική, θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να είναι ενωμένο το Κοινοβούλιο και ότι δεν θα ε, εμφανιστεί ως ένα ψηφοδέες όργανο ενώπιον των ε, διεθνών οικονομικών πιέσεων, των μεγάλων οικονομικών παραγόντων πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω δει πολλές επιχειρήσεις ευρωπαϊκές οι οποίες έχουν αξιοποιήσει πολλά εκατομμύρια από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μέσω των χρηματοδοτήσεων και των επιδοτήσεων και που τώρα θέλουν να αποδυναμώσουν την Ευρώπη γιατί δεν τους συμφέρει. Ε, όχι λοιπόν, αν θέλουμε να ενισχύσουμε την Ευρώπη πρέπει και για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και ιδιαίτερα την ανάπτυξη να δώσουμε ε, χρήματα και βέβαια να επιδείξουμε όσο δυνατόν πιο πολύ ενωτικό πνεύμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Μια διαδικαστική παρατήρηση και πρόταση, γιατί έχουμε και τον Υπουργό ε, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών της Ελλάδας. Έχουμε την ε, Επιτροπή εδώ, τον κύριο Τομάση για να μας δώσει απαντήσεις στο δυνατόν πληρέστερα και γρήγορα όμως, γιατί δεν θέλω να αφήσω τον, τον Υπουργό να περιμένει. Να κλείσουμε έτσι λοιπόν εδώ τον κύκλο των ερωτήσεων. Αν δεν έχετε αντίρρηση, παρακαλώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Τομάση. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλα τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον εισηγητή για τις αξιόλογες προσπάθειες ε, που έχει κάνει σε αυτό το ομολογουμένως ε, πολυσύνθετο ζήτημα που συνδέεται με την πολιτική αλλά και με τις αρχές με τρόπο αρκετά συνήθιστο θα έλεγα. Όταν ε, συμφωνήθηκε το 2008 η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στον τομέα αυτό, ε, υπήρχε πλήρη υποστήριξη από πλευρά ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Πρόκειται για νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε και είναι η μόνη που το επιδιώκει. Θα συμφωνήσω με τους βουλευτές που τόνισαν πόσο σημαντικό είναι να τηρήσουμε τις πολυμερείς διαδικασίες και να τοποθετήσουμε τις ε, διεθνείς διαπραγματεύσεις ε, στο κέντρο των επιδιώξεών μας. Όντως, η συνέλευση της ΣΥΚΑΟ τον Νοέμβρη εστέφθη με επιτυχία ως προς την πρόοδο που ε, σημειώθηκε για μέτρα που εφαρμόζονται σε παγκόσμια κλίμακα. Βλέπουμε ένα μεγάλο αριθμό χωρών που συμφώνησαν ε, για μια παγκόσμια προσπάθεια για το NBN. Είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό το αποτέλεσμα της συνέλευσης του ΙΚΑΟ. Ε, συμφωνήθηκε επίσης ένα διάμεσο μέτρο δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων για τις χώρες που το επιθυμούν ακόμη και πριν το 2020. Μπορεί κάποιοι να ερμηνεύσουν την παράγραφο αυτή του ενδιάμεσου μέτρου ως αμοιβαία συγκατάθεση. Εμείς διαφωνήσαμε και θέσαμε και επιφύλαξη για τη συγκεκριμένη ερμηνεία αυτή της παραγράφου. Θα συνεχίσουμε ε, τις προσπάθειές μας ώστε να καταλήξουμε σε μια συνενετική, θα έλεγα, συμμόρφωση με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα αποφασίσουμε όμως ποιο θα είναι το περιεχόμενο της νομοθεσίας, ε, λαμβάνοντας υπόψη ε, το, τα ευχολόγια των τρίτων χωρών. Ε, στις 16 Οκτωβρίου λάβαμε μια απόφαση ε, που ε, συνιστά και την καλύτερη προσπάθεια που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής για να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις του ΙΚΑΟ. Έχουμε θεσπίσει συγκεκριμένες διατάξεις για τις λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες, για τις πλέον ευάλωτες χώρες και επίσης ε, απηχούν και τις συζητήσεις ε, προ συνελεύσεως και κατά τη διάρκεια της συνέλευσης ε, από μεγάλες χώρες της πολιτικής αεροπορίας και βάσει των προτάσεών τους για τον εναέριο χώρο ή μάλλον προτάσεις που έχουν καταθέσει με γνώμονα τις διατάξεις για τον εναέριο χώρο. Ε, προσδοκώντας την έκβαση της ετήσιας συνέλευσης. Θεωρήσαμε ότι η συρρήκνωση είναι αποδεκτή διότι θεωρούμε ότι θα αρχίσει να λειτουργεί κάποια στιγμή αυτό το παγκόσμιο σύστημα και θέλουμε να μην το υπονομεύσουμε ε, σε αυτό το στάδιο. Ε, ποιο είναι το περιεχόμενο τώρα των διαπραγματεύσεων, ε, τόσο εδώ όσο και στο Συμβούλιο. Ε, περιστρέφονται οι συζητήσει γύρω από τις διάφορες εναλλακτικέ προσεγγίσεις για το μελλοντικό καθεστώς. Υπάρχει η έννοια τη παράταση για την ενδονησιακή κάλυψη μέχρι το 2014. Αυτή είναι η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, έτσι θα έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο για να κάνουμε και τις απαιτούμενες τεχνικές προσαρμόγες ε, για τον εναέριο χώρο. Στη συνέχεια κάποιοι ε, θέλουν να ε, παρατείνουν την παράταση μέχρι το 2026 ε, βάση και των αποφάσεων και των διαδικασιών του ΙΚΑΟ και κάποιοι θεωρούν ότι η παράταση μέχρι το 2020 θα είναι η χρυσή οδός. Πιστεύω ότι πρόκειται για θέματα πολιτικών επιλογών και όλα θα κρυθούν από τις διαπραγματεύσεις. Τα κριτήρια τώρα για να αξιολογήσουμε τις τρεις αναλεκτικές λύσεις θα πρέπει να είναι η απλούστευση, η αηφορία και η σταθερότητα ε, του προγράμματος. Πιστεύουμε ότι η πρότασή μας πληρεί και τα τρία αυτά κριτήρια. Ε, βεβαίως ε, υπάρχει και το θέμα της πολιτικής αποδοχής ε, και το ζήτημα ποιο είναι, σε ποιο σημείο, μέχρι ποιο σημείο θέλουμε να φτάσουμε και τι υποχωρήσεις θέλουμε να κάνουμε. Κάποιοι φορείς, κυρίως οι βιομηχανία, έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για αυτή την προσέγγιση ε, του εναέριου χώρου, αλλά δεν έχουν αντιπροτείνει εναλλακτική η οποία να συνάδει πλήρως με το, τις διατάξεις του ΙΚΑΟ. εμά, ε, νομικός και τεχνικός πώς ε, είναι ε, έγκυρη η πρότασή μας και εξασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους φορείς. Κλείνοντας να σας πω ότι πιέζει πάρα πολύ το χρονοδιάγραμμα και ε, χαιρόμαστε που σημειώνεται η πρόοδος, υπάρχει βούληση για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τρόπο ώστε να βρούμε συγκεκριμένες λύσεις ε, και όχι να αποτελματωθούμε ε, σε συζητήσεις πολιτικού χαρακτήρα, σε συζητήσεις περιαρχών. αρχών. Ας βρούμε τον ταχύτερο δρόμο, τόσο ώστε μέχρι τέλη Απριλίου του τρέχοντος να ολοκληρωθεί η διαδικασία της συναπόφασης. Είναι θαραλέο το εγχείρημα. Πιστεύω όμως ότι είναι εφικτό εάν όλοι λειτουργήσουν καλή την πίστη και κάνουν ε, κάθε δυνατή προσπάθεια. Θα κλείσω με αυτό το μήνυμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω και μια συγκεκριμένη ερώτηση όμως καταθέσει. Ποια είναι τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν μέχρι τώρα εφαρμόσει την ισχύουσα νομοθεσία. Και αν ναι, πώς θα τα αντιμετωπίζετε. Ε, Πρόσωπος της Επιτροπής Πρόεδρε, δεν σκόπευα να αποφύγω την ερώτηση, Νομίζω ότι υπήρχε μια προφορική ερώτηση αργότερα για την εφαρμογή της νομοθεσίας, όπως νομίζετε εσείς. Συνεχίστε, λέει ο Πρόεδρος. Όπως ξέρετε λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το σύστημα των ανταλλαγών εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη. Έχουμε να κάνουμε με την κατανομή αυτή των αρμοδιοτήτων, όπου τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν να ε, κάνουν τις, την ε, εφαρμογή της νομοθεσίας με τις συζητήσεις και την αντιστοίχηση με τους διάφορους ε, φορείς που δυνάμει του ευρωπαϊκού δικαίου φέρουν την υποχρέωση. Η υποχρέωση λοιπόν συμμόρφωσης στο Ευρωπαϊκό Σύστημα ανταλλαγή ε, Εκπομπών ε, στις αεροπορικές μεταφορές ε, παρουσιάζει σημαντικά ποσοστά το 2012. Έχουμε 98% κάλυψη των εκπομπών για το 2012. Ωστόσο έχουμε πρόβλημα η μερική τήρηση, εφαρμογή, πολλές φορές και για πολιτικούς λόγους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τις μόνιμες εγκαταστάσεις έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο διαδικασίες που ποικίλουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο η ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία εξασφαλίζεται από την παρακολούθηση και επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπουμε ότι η πλειονότητα των κρατών μελών είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία. και μπορούμε να εντοπίσουμε τέσσερα διαφορετικά βήματα για την υλοποίηση της οδηγίας. Καταρχάς υπάρχει επίσημη κοινοποίηση, μετά έχουμε, μάλλον την ε, αναγγελία, μετά έχουμε την επίσημη κοινοποίηση της ε, ποινή εφόσον δεν υπάρχει ε, η εφαρμογή και η δυνατότητα της προσφυγής από την αεροπορική εταιρεία όταν, έχουν, όταν έχει ένσταση ως προς τον υπολογισμό των εκπομπών. Και μετά έρχεται η ώρα της κατασταλτικής δράσης και της επιβολής δηλαδή των κυρώσεων. Χρονοδιάγραμμα για αυτά τα στάδια. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να είναι διαφορετικό. Από δύο μέχρι έξι μήνες χονδρικά μπορώ να σας πω. Δεν είναι μια διαδικασία δηλαδή που αρχίζει μια μέρα και την τελειώνει την επομένη. Έχουμε σε όλα αυτά τα στάδια ε, ανάλογα με το, τη γραφειοκρατική επιβάρυνση στο κάθε κράτος διαφορετική διάρκεια των επιμέρους διαδικασιών. Η Επιτροπή λοιπόν εκλήθη από τα κράτη-μέλη να αναλάβει μια συντονιστική δράση, ένα ρόλο διευκόλυνσης, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι, η, ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν την νομοθεσία κατά τρόπο συντονισμένο και ομοιόμορφο. Είχαμε μια πρώτη επιστολή λοιπόν τον Ιούνιο του 2013 που απεστάλλει στις αεροπορικές εκείνες εταιρείε οι οποίες δεν είχαν συμμορφωθεί. Επίσης λέμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε επίπεδο ορμής και ε, επιτάχυνσης των προσπαθειών στην ΙΚΑΟ θα ήταν ακριβώς να έχουμε καλές επιδόσεις ε, στο εσωτερικό μας. Ε, δεν έχουμε καταφέρει 100% αλλά στο επόμενο στάδιο της επιβολής ε, τον Φεβρουάριο θα έχουμε οπωσδήποτε καλύτερα αποτελέσματα. Προς το παρόν δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε την, στρα... την ε, δέσμευση των κρατών μελών στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Εφόσον κάποια καθυστέρηση, ενδεχομένως σύγχυση έχει παρισφρήσει στην εφαρμογή αυτών των διαδικασιών, μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε, να πραγματοποιήσουμε αυτά τα πρώτα βήματα εν ώψη της διαδικασίας παραβιάσεως. Κυρία μου, να σας ρωτήσω για άλλη μια φορά ποια είναι τα κράτη-μέλη, ποια είναι τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν τηρήσει την νομοθεσία, ποια είναι τα κράτη-μέλη και σας ρωτώ για τελευταία φορά. Απάντηση. Δεν υπάρχει κράτος μέλος το οποίο να βρίσκεται σε καθεστώς παραβίασης τη εθνικής του νομοθεσίας ως προς τις δραστηριότητες εφαρμογής και επιβολής. Υπάρχουν διαφορετικά χρονοδιαγράμματα σε διάφορες χώρες. Το χρονοδιάγραμμα που επιτρέπει δηλαδή την ολοκλήρωση των πρώτων επίσημων βημάτων ε, αφορά ένα χρόνο ενδεχομένως ε, ενώ σε κάποιο άλλο κράτος μέλος μπορεί η ποινή να έχει επιβληθεί μέσα στο 12 μήνο και σε κάποιο άλλο οι δραστηριότητες αυτές να εφαρμόζονται κατά διαφορετικό τρόπο. Well, uh, uh, Ας πούμε ότι συμφωνούμε, αλλά όχι και πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι γνωρίζω υπάρχουν επιχειρήσεις από την Κίνα, τη Σαουδική Αραβία και την Ινδία που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που δεν ε, συμμορφώνονται. Και δεν έχουμε αντιδράσει σε αυτή την κατάσταση. Η Air China πετά τακτικά ανάμεσα στην Ελλάδα και το Μόναχο. Η China Eastern κάνει και εσωτερικές πτήσεις στη Γερμανία, Φραγκφούρτη, Αμβούργο. Πιστεύετε ότι υπάρχει τελικά η δυνατότητα να αλλάξουν οι βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις σε σχέση με τις εκπομπές ε, λόγω της πίεσης αυτών των χωρών. Αυτό θα έπρεπε να το επιτρέψουμε. Οι αερομεταφορείς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την δυνατότητα να μη συμμορφώνονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ακόμα και όταν πετούν και δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό των Ευρωπαϊκών Συνόρων. Και αυτό ισχύει και για ε, τις συγκεκριμένες εταιρείες αλλά και για τις χώρες τις οποίες πετούν. Ο κύριος Γκερμπράντι, μία συμπληρωματική ερώτηση. Είπατε και αναφέρθηκα σε αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λέγει ότι δεν υπάρχει εφαρμογή η οποία, η οποία έχει πολιτικά κίνητρα σε ορισμένες χώρες. Ποιες είναι οι χώρες αυτές οι οποίες για πολιτικούς λόγους δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία. Το θέμα δεν είναι αποστολής επιστολής ή οτιδήποτε άλλο, Νομίζω ότι αναφέρθηκα ακριβώς σε αυτά τα οποία είπατε κατά λέξη. Παρακαλώ, ίσως τώρα μπορείτε να απαντήσετε αυτή την τελευταία ερώτηση του κυρίου Γκεμπράντη. Με τα χαράς. Πιστεύω ότι χρησιμοποίησα τη όρους μη συμμόρφωση με πολιτικό κίνητρο. Δεν μιλάμε για μια εφαρμογή, μη συμμόρφωση είπα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει. Αλλά δεν γίνεται ημερών αυτό. Ε, είναι βαρετό και τεχνικό το ζήτημα διότι πρέπει να γίνουν υπολογισμοί των εκπομπών για να ε, διαπιστωθεί η παραβίαση. Μετά χρειάζεται επαλήθευση, ε, μετά ατελείωτη αλληλογραφία ανάμεσα στους φορείς σε τους δικηγόρους τους και τους δικηγόρους των αρμοδίων αρχών. Εγώ σας είπα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί μια συνενετική προσέγγιση για την εφαρμογή σε σχέση με τις εκπομπές για το 2012. Έχουν αποσταλεί επιστολέ κοινοποίηση σε όσους ενδέχεται να έχουν παραβιάσει την ε, νομοθεσία, μεταξύ των οποίων και οι Κινέζοι. Ε, και ε, η διαδικασία συνεχίζεται ανάμεσα στου δικηγόρους των φορέων εκμετάλλευση και τους δικηγόρους των αρμοδίων αρχών. Η συνήθις διαδικασία μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει παραβίαση αυτή καθ' αυτή. Και νομίζω ότι μιλώ εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν σας λέω με πάσα σοβαρότητα δεν θα διστάσουμε να κινήσουμε διαδικασία παραβίασης εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία από πλευράς κάποιου κράτους μέλους. Προς το παρόν δεν έχουν παραβιαστεί ε, σε σχέση με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Καλώς, πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή. Έχω ερωτηματικά, τα οποία μετατρέπονται σε θαυμαστικά ή μάλλον σημεία επισήμανσης και θα ήθελα να ξέρω τι πρόβλημα υπάρχει ως προς την ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών Εάν είναι παραδείγματι, χωρί να ξέρω βέβαια ακριβώ τι συμβαίνει, συμβαίνει στο κάθε κράτο μέλο, εάν η νομοθεσία εθνική δεν επιτρέπει την ταχεία εξέλιξη τη διαδικασία. Ξέρω ότι είναι διαφορετικέ οι πιέσει βεβαίως για ένα κράτο μέλο εάν το παρακολουθεί κάποιο και του λέει προχώρη πιο γρήγορα από ότι αν δεν επέμβουμε. Ε, δεν είναι καθόλου ικανοποιητική η κατάσταση. Σα μεταφέρω τουλάχιστον και παρακαλώ να μεταφέρετε και εσεί από πλευρά σε αυτό το μήνυμα. Δεν είναι ικανοποιητική η κατάσταση και δεν μπορεί να παραμείνει η κατάσταση όπω έχει. Ευχαριστώ και ο εισηγητή. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους είναι πολύ πιο σαφής η υποστήριξη που εκδηλώνεται σήμερα, εκτός από το ECR. Οι πράσινοι ξέρουμε ότι θέλουν να πάνε πιο πολύ στα άκρα. Ε, εν γέννη όμως όλοι είμαστε υπέρ της διατήρησης αυτής της προσέγγισης και για το αερέριες μεταφορές. Για να συνοψίσω. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτελέσει πιο αποτελεσματικά το ρόλο του θεματοφύλακα. Και ενώ η κατάσταση μπορεί να είναι διαφορετική από ό,τι είχαμε την εντύπωση και, δεν υπάρχουν, ε, και αν δεν υπάρξουν προβλήματα, τότε πάμε στον τριμερή διάλογο και διευκρινίζουμε την κατάσταση. Εάν όμω πρέπει να περάσουν τρία χρόνια μέχρι να επιβληθούν κυρώσει, τότε αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συστήσουμε στον τριμερή διάλογο και να είμαστε και πιο σαφεί στι διατυπώσει που θα επιλέξουμε. Εγώ δεν είμαι πάντω διατεθειμένο να κλείσω τριμερή διάλογο όταν δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία. Με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεν μεριμνούν επαρκώς. Έχω μιλήσει με τον Γάλλο Υπουργό Περιβάλλοντος, ο οποίος ε, μου εξήγησε διαμακρών και ε, γιατί πρέπει να εφαρμοστεί το stop the clock. Όταν όμως ε, τον ρώτησα γιατί η Γαλλία δεν εφαρμόζει το δίκαιο, μου λέει «Α, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι υπουργός μεταφορών, είμαι μόνο περιβάλλοντος» και όταν ξέρουμε τι είδους προτεραιότητα είναι το να θυμίσουμε και στους Κινέζους ότι έχουν να τηρήσουν μια συγκεκριμένη νομοθεσία, πράγμα το οποίο κανείς δεν κάνει. Αυτό θα το πω στον Έλληνα Υπουργό. Στην κατάσταση αυτή εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να κλείσω το τριμερή διάλογο. Απέστειλα πέρσι ήδη επιστολή στην Λιθουανική Προεδρία. Ούτε απάντηση δεν μου δώσανε. Ούτε από το προσωπικό του Συμβουλίου, ούτε από το προσωπικό της Επιτροπής. Με ρίμνησε κανείς να μου δώσει μια απάντηση για το εάν και από ποιου εφαρμόζεται ικανοποιητικά νομοθεσία. Με αυτού του όρου δεν κλείνω ο τριμερή διάλογο λοιπόν. Και έτσι, τελευταίο θέμα, το 2007-2008 ούτε η Επιτροπή ήταν ούτε το Κοινοβούλιο αυτοί που επέβαλαν, όπως στην πραγματικότητα το έκανε το Συμβούλιο δηλαδή, επέβαλαν τη δυνατότητα για μια χώρα τρίτου, για μια αεροπορική εταιρεία τρίτου κράτους να μπορεί να εφαρμόζει, να επιβάλλεται μάλλον να εφαρμόζει το σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θυμίσω σε ορισμένους ότι δεν ήταν θέση Επιτροπή, το Συμβούλιο ενέγραψε αυτή την διάταξη μέσα στον ε, στο νομοθέτημα, στην οδηγία. Αυτό λοιπόν πρέπει να το υπενθυμίσουμε στην επιστολή που θα στείλουμε ε, και δεν μπορεί να μην εφαρμόζεται οδηγία και νομοθεσία που ισχύει. Τελευταία παρατήρηση, η επόμενη παρατήρηση καλύτερα, η κυρία Φώστερ μας είπε δεν είναι δογματικές θέσεις Χαίρομαι που είναι πάντα τόσο οι τοποθετήσεις απέναντί μου, όπου μου δείχνει ότι πάντα ο κακός ε, της υπόθεσης είναι η Επιτροπή. Όχι, ο κακός της υπόθεσης δεν είναι η Επιτροπή, η Επιτροπή είναι πάντα πολύ ευέλικτη και είναι διτεθειμένη να καταλήξει μια ρεαλιστική, πραγματιστική θέση. Ο μεγάλος όμως ε, των δογματικών θέσεων ονομάζεται George Osborne ε, ανήκει στη Βρετανική κυβέρνηση, είναι υπουργό των οικονομικών, λέει «Α, εγώ δεν συζητώ τέτοια θέματα», ούτε ένα λεπτό ούτε μισή λίρα δεν στέλνω στην Ευρώπη και έτσι οποιοδήποτε επιβάτης ταξιδεύει από το Λονδίνο στη Σανχάη ή πιο πέρα και με business και με δεν ξέρω τι δεν... Μα έτσι είναι, μα έτσι είναι, δεν πληρώνει. Ε, άκουσε να σου πω Τζάκη, δεν μπορεί να μου λες ότι δεν συμβαίνει αυτό που ισχύει. Πρόκειται για ένα φόρο 200 ευρώ. Για λόγους δογματικούς που επιβάλλει η Βρετανική κυβέρνηση. Το οποίο, ο οποίος φόρος, το οποίο τέλος μας γεννά πολλά προβλήματα. Τελευταία παρατήρηση, η Ήτρε, μόλις ψήφισε από ό,τι έμαθα. Ενέκρινε λοιπόν 29 22, 3, 29 υπέρ, 22 κατά 2 αποχές. Ενέκρινε, είναι πολύ στενά όμως τα περιθώρια. Άρα είναι πολύ αυτοί στην Ήτρο που προτιμούν την πρόταση airspace. Εάν θυμηθούμε την απόρριψη από την Ήτρε του backloading ε, και την ανατροπή αυτού του αποτελέσματος από την Ολομέλεια πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα της Ήτρε δεν αποτελεί απόδειξη ότι το θέμα του ενέργειου χώρου την χάνει επαρκούς υποστήριξης. Την επόμενη εβδομάδα θα το ψηφίσουμε εμείς, θα δούμε. Και πρέπει να δούμε επίσης αν εξασφαλιστεί συμβιβαστική λύση. Αυτό εμένα πολύ θα με χαροποιούσε. Εάν όμως δεν τα καταφέρουμε, πρέπει να γίνει την επόμενη εβδομάδα ψηφοφορία. Και πιστεύω ότι θα έχουμε υποστήριξη για την πρόταση της Επιτροπής, τροποποιημένη. Ευχαριστώ. Ε, έχουμε τον Υπουργό στην πόρτα και περιμένει. Θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα. 30 Ιανουαρίου είναι η ψηφοφορία. Και της εντολής. αν τα καταφέρουμε τον Απρίλιο 2014 στην Ολομέλεια, μπορεί να έχουμε μια ευκαιρία να κλείσουμε το θέμα. Αλλά ήθελα ήδη να πω ότι αισθάνομαι δυσφορία και αρκετέ αμφιβολίε για το κατά πόσον δεδομένη τη στάση τη Επιτροπή και των απαντήσεων που δεν έδωσε ε, μπορεί να προχωρήσει το θέμα αυτό. Α περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη.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 εδώ τον εκπρόσωπο της Προεδρίας του Συμβουλίου, Πρόεδρο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Ο προσκεκλημένος μας κύριος Γιάννης Μανιάτης είναι εδώ. Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε εδώ. Έχετε το λόγο βεβαίως ως προσκεκλημένος πρώτος για να μας παρουσιάσετε τα κύρια σημεία της Προεδρίας σας και Μετά θα λάβει χώρα μια ε, σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων με τους συντονιστές που θα ακολουθήσει και ένας γύρος ερωτήσεων με τους λοιπούς συναδέλφους. Παρακαλώ δε τους συντονιστές να είναι στο δυνατόν σύντομες ερωτήσεις για να έχουν όλη την ευκαιρία να ε, διατυπώσουν τις δικές τους ερωτήσεις. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, ε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να είμαι σήμερα μαζί σα και να σα παρουσιάσω τι προτεραιότητε της Ελληνική Προεδρίας. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω υπενθυμίζοντα αυτά που είπε ο Έλληνα Πρωθυπουργό στο Στρασβούργο και τα οποία αφορούν τι ευχαριστίες που θέλουμε να απευθύνουμε εκ μέρου του ελληνικού λαού προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι στάθηκε δίπλα στον ελληνικό λαό και τις θυσίες που υφίσταται το τελευταίο χρονικό διάστημα και χαιρόμαστε γιατί πραγματικά η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών έχει αναγνωρίσει τις θυσίες του ελληνικού λαού και εμείς δεν θα το ξεχάσουμε. Πριν σας ε, κάνω μια ειδικότερη αναφορά στα ζητήματα της, των προτεραιοτήτων για τα θέματα του περιβάλλοντος, επιτρέψτε μου πολύ συνοπτικά σε τίτλους να δώσω τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες συνολικά της ελληνικής προεδρίας. Ο πρώτος στόχος είναι η αποτελεσματική εφαρμογή και προώθηση του Συμφώνου Ανάπτυξης και Απασχόλησης με τελικό στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της ανεργίας και ιδιαίτερα του προβλήματος της ανεργίας των νέων. Η δεύτερη προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας είναι η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης με ιδιαίτερη έμφαση στις διαπραγματεύσεις για την τραπεζική ενοποίηση. Η τρίτη προτεραιότητα αφορά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη στήριξη της κινητικότητας. Τέλος, και αυτή η τέταρτη προτεραιότητα έχει άμεση σχέση με τη δική μας Επιτροπή, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, η ελληνική Προεδρία φιλοδοξεί να εισαγάγει μια νέα οριζόντια πολιτική για τις θαλάσσιες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό φιλοδοξούμε να ανασχεδιάσουμε τη θαλάσσια πολιτική με ορίζοντα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2014. Στόχος μας είναι να συμπεριληφθούν σε αυτή θέματα όπως το περιβάλλον, η αλληλεία, η ενέργεια, οι θαλάσσιες μεταφορές, ο τουρισμός, η ασφάλεια, και ασφαλώς οι περιφερειακές στρατηγικές για επιμέρους θαλάσσιες περιοχές της Ένωσης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο, που σε συνεργασία της τωρινής ελληνικής προεδρίας και της επόμενης Ιταλικής προεδρίας πιστεύουμε ότι θα οριμάσουν αρκετά. Επιτρέψτε μου επίσης να σημειώσω πως ε, από την θέση της Προεδρίας θέλω να τονίσω την ιδιαίτερη σημασία που έχει η Επιτροπή σας στο πολιτικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό γίγνεσθε της Ευρώπης, διότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος θεωρείται από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες ως μια ασφαλιστική δικλίδα για να προωθήσουμε τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τον πλανήτη, που είναι το ζήτημα ασφαλώς της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος. Έτσι, εκ μέρους και της Προεδρίας, θέλω να ζητήσω να έχουμε την στήριξή σας και τη βοήθειά σας κατά τη διάρκεια του σύντομου χρονικού διαστήματος της Προεδρίας, γιατί πράγματι πιστεύουμε πως η στενή συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και το Συμβούλιο ε, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής θα μας βοηθήσει να επισπεύσουμε την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Σημειώνω ορισμένες πολύ βασικές παρατηρήσεις που τις γνωρίζουμε όλοι, αλλά θεωρώ χρήσιμο σε μια τέτοια πολύ σημαντική ε, στιγμή για μας ως Προεδρία απέναντί σας να τα ξαναφέρω στο μυαλό μας. Πρώτον, δυστυχώς δεν έχει πετύχει η ανθρωπότητα μέχρι σήμερα το βασικό της στόχο να πηγαίνουμε προς μια αύξηση της παγκόσμιας θερμότητας κάτω από τους δύο βαθμούς Κελσίου. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, άρα πρέπει συνολικά η ανθρωπότητα να λάβει ακόμα πιο ε, αποτελεσματικά μέτρα ώστε να, να μειωθεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας και αυτό είναι το νόημα και το βασικό συμπέρασμα της τελευταίας αναφοράς των Ηνωμένων Εθνών για το GAP Report. Η δεύτερη παρατήρηση είναι πως οι αναπτυσσόμενες χώρες παράγουν το περίπου 60% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση να παράγει μόλις το 11%. Η τρίτη θετική παρατήρηση και έχει να κάνει με αυτό που ως Ευρωπαίοι πολίτες νομίζω μπορούμε να λέμε ε, σε όλους τους υπόλοιπους συνανθρώπους μας είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη περιοχή στον κόσμο που έχει εντάξει στο συνολικό της προϋπολογισμό ένα κονδύλι της τάξης των 180 δισεκατομμυρίων ευρώ για όλες τις οριζόντιες πολιτικές εν ώψη της προγραμματικής περίοδου 2014-2020 έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής. Η τέταρτη παρατήρηση σχετίζεται με το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που αναφέρει ότι αν δεν προσέξουμε την βιοπικιλότητα τότε χάνουμε ήδη περίπου 3% από το παγκόσμιο καθάριστο εγχώριο προϊόν. Και έχει μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα σε οικονομικούς αναλυτές, να τονίζουμε από όλες τις πλευρές τη σπουδαιότητα της βιοπικιλότητας. Αυτές οι δράσεις στοιχίζουν πάνω από 450 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Και τέλος να θυμίσω αυτό που και από την πλευρά της ενέργειας, του Συμβουλίου Ενέργειας πρέπει να είναι κατανοητό, ότι ζούμε σε έναν πλανήτη όπου 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπων δεν έχουν ηλεκτρισμό και περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπων δεν έχουν στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής για να μαγειρέψουν το καθημερινό τους φαγητό. Μετά από αυτές τις πολύ σύντομες παρατηρήσεις, επιτρέψτε μου να έρθω όσο μπορώ πιο σύντομα στις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας. Η επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση είναι ένας στόχος μας για την πρόταση για τη μεταφορά αποβλήτων και την πρόταση για ένταξη της αεροπλοείας στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Ως προς την πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού της μεταφοράς αποβλήτων, η προσπάθεια για επίτευξη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση υποστηρίζεται σχεδόν από το σύνολο των καρτών μελών πιστεύουμε ότι με τη δημιουργική συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία θα είναι η καλύτερη δυνατή για όλους. Για το θέμα της αεροπλοείας, ένα πολύ σημαντικό θέμα, γνωρίζουμε τη σημασία της πρότασης για τη διασφάλιση ενός σταθερού νομικού περιβάλλοντος χωρίς ασάφειες για τις αεροπορικές εταιρείες. Επίσης γνωρίζουμε πόσο σημαντική επίδραση θα έχει η απόφαση που θα πάρει η Διεθνής Ένωση της Αεροπλοείας, ο ΑΙΚΑΟ, και στις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας το 2006 έτσι ώστε στο τέλος της ημέρας να έχουμε ένα μέτρο που θα βασίζεται, ένα παγκόσμιο μέτρο που θα βασίζεται στη λειτουργία της αγοράς. Αναγνωρίζουμε και σημειώνουμε <clears throat> ότι για λόγους πολιτικής αξιοπιστίας της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απόλυτη ανάγκη να εξασφαλίσουμε άμεσα μια συμφωνία στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Έχοντας αυτά υπόψη, Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε επικοδομητικά με την Επιτροπή σας με σκοπό να πετύχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Στα δύο προηγούμενα, στις δύο προηγούμενες προτάσεις πρέπει να προσθέσουμε την πρόταση του κανονισμού για τα ξενικά χωροκατακτητικά είδη. Για την πρόταση αυτή είχε υπάρξει από την αρχή μια συγκρατημένη αισιοδοξία για να επιτευχθεί συμφωνία λόγω ακριβώς του περιορισμένου χρονικού διαστήματος που έχουμε στη διάθεσή μας χάρη όμως την πρωτοβουλία του Ευρωκοινοβουλίου να επισπεύσει κατά δύο εβδομάδες περίπου την ψήφιση της πρόταση κανονισμού στην Επιτροπή σας, σε συνδυασμό με την πρόοδο που σημειώθηκε κατά το τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών, μπορεί κανείς να θεωρήσει και το θεωρεί αυτό η Προεδρία ότι έχουμε σημαντικές πιθανότητες να πετύχουμε τελική συμφωνία. Σημειώνω ότι ασφαλώς υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα, σημαντικές ακόμη διαφωνίες, ανάμεσα στα διαφορετικά κράτη-μέλη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την συμπερίληψη ή όχι ειδών που προέρχονται από τις ίδιες τις χώρες της Ένωσης στον κατάλογο ξενικών χωροκατακτητικών ειδών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Και βεβαίως ένα άλλο θέμα που απασχολεί είναι το εύρος των εξαιρέσεων μετά από άδειε που μπορούν να δίνονται υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και αρκετά σημεία σύγκλησης. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο στο συγκεκριμένο θέμα γιατί είμαστε σε πλήρη εξέλιξη της συγκεκριμένης διαπραγμάτευσης αλλά θέλω πραγματικά να ελπίζω ότι σε δύο με τρεις μήνες από σήμερα θα καταφέρουμε όλοι μαζί Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και ασφαλώς Επιτροπή να χαιρετήσουμε την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα μας επιτρέψει για πρώτη φορά να έχουμε ένα αυστηρό νομικό, νομοθετικό και αποτελεσματικό πλαίσιο για να προστατεύσουμε την βιοπικιλότητα στα κράτη-μέλη. Μια σημαντική προτεραιότητα της Προεδρίας μας είναι ασφαλώς η συζήτηση και η προώθηση της χθεσινής, του κειμένου της χθεσινής ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πακέτο κλίμα, κλιματική αλλαγή, ενέργεια μπροστά στο 2030. Και να σημειώσω ότι αφορά πολύ σημαντικές αποφάσεις που σχετίζονται με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα και της ενέργειας αλλά και στον τομέα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Για το λόγο αυτό άλλωστε το θέμα θα απασχολήσει τις ομάδες περιβάλλοντος και ενέργειας του Συμβουλίου έτσι ώστε να υπάρξει μια ουσιώδης ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Υπουργών στα αντίστοιχα συμβούλια που θα γίνουν μέσα στο Μάρτιο. Λόγω της σημασίας του θέματος, το συγκεκριμένο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και της ενέργειας θα συζητηθεί και στο Συμβούλιο Κορυφής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο τέλη Μαρτίου. Η προοπτική είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές συζητήσεις ανάμεσα σε όλους τους εταίρους, Συμβούλιο, Επιτροπή, ε, Κοινοβούλιο, να έχουν ολοκληρωθεί σχετικές συζητήσεις μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Να έχει ολοκληρωθεί δηλαδή η συζήτηση με την ολοκλήρωση και της επερχόμενης Ιταλικής Προεδρίας. Θέλω να σημειώσω αυτά που ανέφερε χθε ο πρόεδρος Μπαρόζο στη δήλωσή του κατά την ανακοίνωση του κειμένου, ότι δηλαδή η δράση για το κλίμα είναι κεντρική σημασία για το μέλλον του πλανήτη μας, ενώ μια πραγματικά ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική μπορεί να είναι το κλειδί και για την ανταγωνιστικότητά μας. Θεωρώ λοιπόν πως η χθεσινή δέσμη μέτρων μπορεί να αποτελέσει ένα αρκετά ρεαλιστικό πλαίσιο συζήτησης διαλόγου για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση των δύο θεμάτων της κλιματικής αλλαγής και της ενέργειας. Η στόχοι που θα πρέπει και η Προεδρία να έχει στο μυαλό της και όλοι μας εν ώψη της συζήτησης που θα ανοίξει, και έχει ήδη ανοίξει από χθε, είναι η ακόλουθη. Πρώτον, προβλεψιμότητα και σιγουριά στα κράτη-μέλη και τους επενδυτές για το τι θέλουμε να κάνουμε ως Ένωση μέχρι το 2030. Δεύτερον, η λήψη κοινή ευρωπαϊκή θέση για τι δεσμεύσει μειώσεων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εν ώψη τη αναμενόμενη και ελπίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί παγκόσμια συμφωνία για τι εκπομπέ αερίων το 2015 στο Παρίσι. Η τρίτη επιλογή είναι να υπάρχει ασφάλεια ενεργειακής προσφοράς μέσα από την ανάπτυξη της ενεργειακής εξοικονόμησης και της ενεργειακής αποδοτικότητας, αλλά και μέσα από την ανάπτυξη και βελτίωση δικτύων ενεργειακής υποστήριξης, τα λεγόμενα PCI, τα προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Και βεβαίως η ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλού άνθρακα που θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας και θα προωθήσουν την έρευνα και την καινοτομία. Πιστεύουμε ως Προεδρία ότι είναι προς το συμφέρον όλων των λαών της Ένωσης να οικοδομήσουμε μια οικονομία που θα διατηρεί τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και θα δημιουργεί και νέες, ενώ ταυτόχρονα θα είναι λιγότερο εξαρτημένη από εισαγωγές ενεργειακών αγαθών εκτός Ευρώπης και θα στηρίζεται πολύ περισσότερο στην εγχώρια παραγωγή καθαρής ενέργειας. Δεν θα επεκταθώ στις επιμέρους ε, παραμέτρους του συγκεκριμένου πακέτου, θέλω όμως να επισημάνω ότι είναι πραγματικά θετικός και φιλόδοξος ο στόχος για την ε, μείωση των εκπομπών κατά 40% μέχρι το 2030 σε σχέση με το έτος αναφοράς 1990 και αυτός είναι ένας οικονομικά αποδοτικός στόχος στην πορεία προς μια ευρωπαϊκή οικονομία χαμηλών εκπομπών ε, ε, χαμηλού άνθρακα και είναι γνωστό σε όλους μας ότι το Κοινοβούλιο έχει βοηθήσει αποφασιστικά στο να περάσουν, να προωθούν τέτοιου είδους θέσεις. Και ασφαλώς να θυμίσω ότι η Ένωση, η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να έχει έναν πολύ ισχυρό προσανατολισμό στα ζητήματα της εισαγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο όλων των κρατών μελών και βεβαίως περιτεύει να σημειώσω την μεγάλη σπουδιότητα της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Να σας διαβεβαιώσω ότι η Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διευκολύνουμε τις συζητήσεις εντός του Συμβουλίου για το θέμα αυτό, ενώ επίσης θα προωθήσουμε όσο είναι δυνατόν τις συζητήσεις για τις νομοθετικές αλλαγές, για τις δομικές αλλαγές που χρειάζεται να κάνουμε στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων. Περνώντας τώρα σε ένα άλλο θέμα, τις εκπομπές ναυτιλίας, να σημειώσω ότι σκοπός μας είναι, αν και ο χρόνος δεν βοηθάει τόσο πολύ σε αυτήν την κατεύθυνση, να προωθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το συγκεκριμένο θέμα για την παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών της ναυτιλίας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο τεχνικό θέμα, το οποίο αναμένεται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά και σχετίζεται με την εφαρμογή του και σε πλοία τρίτων χωρών. Κατά συνέπεια, έχουμε βαθιά ανάγκη ο κανονισμός που θα υιοθετηθεί να είναι λειτουργικός, να μην δημιουργεί προβλήματα εφαρμογής, ενώ ταυτόχρονα να λάβουμε πρόνοια ώστε να ελαφρυνθούν όλα τα πιθανά διοικητικά ε, βάρη και το άχθος. Θέλουμε επίσης να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο στις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο πακέτο για την επικύρωση της τροποποίησης της Ντόχα. Αναγνωρίζουμε ότι η όσο το δυνατόν ταχύτερη επικύρωση είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ένωση ενώ των διεθνών διαπραγματεύσεων ε, μπροστά στο Παρίσι το 2015 παρά τους χρονικούς περιορισμούς επίσης που υπάρχουν θα επιδιώξουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Σημειώνω επίσης τις προτεραιότητες που έχουμε αναφορικά με το πακέτο για την ποιότητα του αέρα και εδώ αναφέρομαι στις επιδιώξεις μας να προχωρήσουμε και τις τρεις νομοθετικές προτάσεις που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή την αναθεώρηση της οδηγίας για τα National Emission Ceilings, τα NEC, τη νέα πρόταση οδηγίας για τις εγκαταστάσεις καύσης μεσαίου μεγέθους και την αναθεώρηση και την επικύρωση του αναθεωρημένου πρωτοκόλλου του Γκέτεμπουργκ. Σκοπεύουμε μάλιστα τον Ιούνιο να έχουμε την ευκαιρία για μια ουσιαστική συζήτηση για τα θέματα αυτά στο Συμβούλιο Υπουργών. Το θέμα τώρα της πλαστικής σακούλας, των πλαστικών σακουλών, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι πλαστικές σακούλες συσσωρεύονται στο περιβάλλον, ειδικά με τη μορφή θαλάσσιων αποβλήτων, με τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το Συμβούλιο έχει ήδη αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα αυτού του θέματος και θα επιδιώξουμε την μέγιστη δυνατή ορίμανση του συγκεκριμένου θέματος. Τώρα, περνώντας στα μη νομοθετικά ζητήματα, θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά και επιλεκτικά τα ακόλουθα. Πρώτον, τη συνεισφορά του Συμβουλίου Περιβάλλοντος στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, θέμα το οποίο θα συζητήσουμε στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος το Μάρτιο. Δεύτερον, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη βιοπικιλότητα εν ώψη της διεθνούς διάσκεψης το COP12 στην Κορέα για την βιοπικιλότητα τα συμπεράσματα αυτά θα πρέπει να τα υιοθετήσουμε στο Συμβούλιο Υπουργών του Ιουνίου. Τρίτον, το συντονισμό της Ένωσης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης αναφορικά με το Ρίο Plus Έντι, και την προετοιμασία των κοινοτικών θέσεων εν της συνάντησης των Ηνωμένων Εθνών στο Ναϊρόμπι τον Ιούνιο. Τέταρτον, την προετοιμασία και προώθηση των θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήματα των διεθνών συμβάσεων, όπως είναι η Σύμβαση του Άρχους και η Σύμβαση ΕΣΠΟ. Επίσης, προτεραιότητά μας είναι η ορίμανση των θέσεων της Ένωσης εν ώψη πάντα της αναμενόμενης παγκόσμιας διάσκεψης στο ε, Παρίσι για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις που θα έχουμε τον Ιούνιο στη Βόνη και στη συνέχεια την παγκόσμια διάσκεψη στη Λίμα το COP20 στο τέλος του 2014 και πιθανόν γι' αυτό το λόγο να έχουμε υπουργικέ συνεδριάσεις στη Βόνη με σκοπό να διευκρινίσουμε συγκεκριμένα θέματα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της παγκόσμιας διάσκεψης και Λίμα. Να σας ενημερώσω επίσης κύριοι Ευρωβουλευτές ότι στις 14 και 15 Μαΐου 2014 θα γίνει το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος στην Αθήνα με βασικό θέμα τη γαλάζια ανάπτυξη. Η γαλάζια οικονομία στην Ένωση προσφέρει δουλειά σε πάνω από 5 εκατομμύρια ανθρώπους και συνεισφέρει με περίπου 500 δισεκατομμύρια ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία. Στόχος της Προεδρίας, στόχος της Ένωσης είναι η προώθηση του ζητήματος της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης της γαλάζιας ανάπτυξης, έτσι ώστε μέχρι το 2020 να έχουμε 7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και περίπου συνεισφορά 600 δισεκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία. Μάλιστα, σε συνεργασία με την επερχόμενη Ιταλική Προεδρία, έχουμε ονομάσει το 2014 ως έτος της Μεσογείου και γι' αυτό θα οργανώσουμε μια υπουργική διάσκεψη με θέμα το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν και αυτά τα θέματα. Τέλος, ολοκληρώνοντας την παρουσίασή μου και ευχαριστώντας για την προσοχή σας και την κατανόησή σας, να πω ότι το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει δύο φορές κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, στις 3 Μαρτίου στις Βρυξέλλες και στις 12 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θέλω να καλέσω για άλλη μια φορά να σας καλέσω να μας βοηθήσετε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Εμείς ως Προεδρία θα επιδιώξουμε την ως το δυνατόν πιο δημιουργική συνεργασία με την Επιτροπή σας και να επαναλάβω για άλλη μια φορά πως χαιρόμαστε που έχουμε μια σύνθεση Επιτροπής Επιτροπής Περιβάλλοντος που βοηθά αποφασιστικά τους Ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να συμβάλλουν στην επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Υπουργέ. Πολλή δουλειά έχετε να αναλάβει. Ο ε, δικός μας χρόνος τελειώνει βέβαια γιατί μέχρι, μέχρι το Πάσχα πρέπει λίγο πολύ να έχουμε τελειώσει τη δουλειά μας. Το κοινοβούλιο έχει μόνο τέσσερις μήνες και de facto τρεις θα λέγαμε περιθώριο, αλλά θα τα καταφέρουμε ελπίζουμε μαζί και βλέπω ότι έχουμε επισκέψεις. Σημαντικές προσωπικότητες από τη Γαλλία. Εκείνοι οι οποίοι ε, είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου όπως το εφαρμόζουμε εμείς στο κάθε διαμέρισμα της Γαλλίας, οι νομάρχες δηλαδή, είναι εδώ παρόντες, 8 νομάρχες και τους καλωσορίζουμε θερμά. Genau, da hinten Gut, dann steigen wir ein in die Runde. In... Ξεκινάμε λοιπόν τώρα με τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Πρώτα τους συντονιστές. Ο κύριος Πετερλής είναι πρώτος, οι λοιποί συνάδελφοι με τη σειρά τους. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για τις ε, παρουσία σα. Θα ήθελα ρητά να εκφράσω την αλληλεγγύη μου με τον κόσμο στην Ελλάδα που έχει κάνει τόσες θυσίες. Είχαμε και τον συνάδελφό σας Υπουργό Ενέργειας ε, ακόμη και θέλαμε να πούμε πόσο ε, σημαντικό, στο δημόσια υγεία και πόσο σημαντικό είναι το να υπάρχει αυτή η υποστήριξη. Υποστήριξη και αλληλεγγύη που ούτε να φανταστούν οι Αμερικανοί Φερρυπίν δεν θα μπορούσαν ε, να ε, δεν θα μπορούσαν στα όνειρά τους. Γι' αυτό για να απαντήσουμε σε διάφορα ψέματα που διαδίδονται. Επίσης, η Πορτογαλία η οποία έχει επίσης να αντιμετωπίσει δύσκολα προβλήματα στο θέμα της ε, ενέργειας και που είδαμε πολύ σημαντικά προγράμματα από τον κύριο Μορέρα Ελπίζουμε μετά το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο κατάφερε η Ελλάδα κατά τρόπο φαινομενικό, κατά τρόπο εντυπωσιακό πραγματικά, να μπορέσουν και εκείνοι με τις προτάσεις Μορέρα να προχωρήσουν. Θα έχουμε τριμερή διάλογο. Ε, μας απασχόλησε το θέμα των εκπομπών. Ε, μόλις τώρα θα το δούμε. Μάλλον θα, θα δούμε μια αντιπαράθεση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό. Και θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε, όπως είπαμε και μεταξύ μας, ότι τα ε, κράτη-μέλη εφαρμόζουν την νομοθεσία όπως έχει συμφωνηθεί. Το ένα έτος αυτό του Stop the Clock, ε, διότι υπάρχουν εταιρείες αεροπορικές οι οποίες ε, πετούν στα κράτη-μέλη από την Αθήνα στο Μόναχο Φερρυπίν και δεν επιτρέπεται να μην εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο. Στον τριμερή διάλογο λοιπόν θα σας παρακαλέσω το ταχύτερο δυνατό πιο σε όσο πιο πρώιμο στάδιο της διαδικασίας να στραφείτε σε εμάς, ε, να στραφείτε σε εμάς για να μας ενημερώσετε, αλλά να προσπαθήσετε να πείστε και τους συναδέλφους σας και τους υπουργούς των οικονομικών στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε τα μέτρα που θα υιοθετούνται να είναι στο δυνατόν πιο εστιασμένα και να έχουμε μεγαλύτερη αποδοχή για τα προγράμματα έρευνας για την κλιματική πολιτική. Μέχρι τώρα ξέρουμε ότι οι Υπουργοί των Οικονομικών ιδιαίτερως είναι ε, ακολουθούν πολύ δογματικές θέσεις ε, και δεν μετακινούνται καθόλου από τις θέσεις τους. Ε, επίσης, χθες συζητήθηκαν οι στόχοι του 2030 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να τους συζητήσουμε διεξοδικά, αλλά θα ήθελα να σας καλέσω να ρίξετε μια ματιά στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς στο μέλλον και πώς, μπορεί το ευρωπαϊκό, ε, πώς μπορούν οι στόχοι αυτοί να μεταφραστούν σε ευρωπαϊκό δίκαιο. Μας ε, περιέγραψε ένα ρόθινο πίνακα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα για την ενέργεια, ενώ το ζήτημα της διακυβέρνησης, των governance, δεν έχει ακόμα κλείσει. Εμείς ως Κοινοβούλιο αυτό το θεωρούμε κήρυξη πολέμου. Δεν μπορούμε δηλαδή να προχωρήσουμε, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Επιτροπή και εφόσον υπάρχει μια πρόταση η οποία παρεμβαίνει στις ε, αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, δεν το δεχόμαστε μέσα σε ένα δημοκρατικό σύστημα. Η Ελλάδα είναι η μητέρα της δημοκρατίας. Γι' αυτό λοιπόν και πρέπει ό,τι κάνουμε να προχωρεί μέσα από την συναπόφαση με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και με καμία άλλη μορφή διακυβέρνησης, governance. Ευχαριστώ πολύ τον Πέτερ Λίσε. Παρακαλώ να είστε όλοι πολύ σύντομοι, παρακαλώ. Κυρία Μακέβαν. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ξέρω ότι καλείστε να κλείσετε κάποια θέματα πριν τις εκλογές, κάτι το οποίο δεν θα είναι εύκολο πριν και από, την, ε, τον τερματισμό της κοινοβουλευτικής περίοδου. Όπως είπατε, έχουμε μπροστά μας ε, το πακέτο 2030. Κάποιοι από εμά πιστεύουν ότι το πακέτο αυτό δεν είναι πολύ φιλόδοξο. Αν συγκρίνω το που είμαστε σήμερα και πού βρισκόμασταν το 2009 όταν ο Έλληνας τότε επίτροπος, ο κύριος Δήμας, είχε ε, δημιουργήσει ένα πακέτο για το κλίμα πάρα πολύ φιλόδοξο που έδιδε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ηγέτιδα θέση. Αντίθετα αυτό το οποίο μας παρουσίασε χθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία σχέση. Είναι μια υπαναχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα. Δεν κατηγορώ την Επίτροπο, αλλά η Επιτροπή γενικά δεν έχει πολιτική βούληση και στην ουσία οι Επίτροποι που ασχολούνται με θέματα οικονομίας και βιομηχανίας κυριαρχούν πλέον. Εμείς ψηφίσαμε τρεις βασικούς στόχους για το 2030 πριν μερικές εβδομάδες. Δεν βλέπω πώς θα μπορέσουμε εμείς να έχουμε μια ισχυρή βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς αυτούς τους στόχους. Οι στόχοι δεν έχουν σημασία. Σημασία έχουν τα μέσα για την επίτευξή τους. Ελπίζω να χρησιμοποιήσετε λοιπόν την Προεδρία σας, να μην είστε υποχωρητικός. Έχουμε το 2015 πράγματι τη συνάντηση στο Παρίσι, αλλά δεν έχουμε καμία ηγετική πρωτοβουλία ως προς αυτό. Δεύτερο κάτι το οποίο, για το οποίο δεν είστε υπεύθυνο, αλλά σαν Συμβούλιο πρέπει να το γνωρίζετε. Πρόκειται για τους ε, ενδοκρινικούς αναστολής, πρόκειται δηλαδή για χημικές ουσίες οι οποίες έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ξέρετε ότι απαγορεύτηκε το μπιτφενόλι 1 ή μπιτφενόλι α για την κατασκευή πλαστικών σκευών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υποσχέθηκε ότι θα υπήρχε δράση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τους ενδοκρινικούς αναστολής. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο και υπάρχει μια περαιτέρω ετήσια καθυστέρηση. Για μια ακόμη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχωρεί και είναι αδύναμη στις πιέσεις του βιομηχανικών λόμπι. Είστε πολιτικός και εγώ είμαι πολιτικός. Πράγματι θα πρέπει να είμαστε γενναίοι μερικές φορές γιατί αλλιώς τίποτα δεν θα αλλάξει και θα χειροτερεύσουν τα πράγματα. Παρακαλώ εξετάστε το θέμα των αναστολέων αυτών. Υπάρχει ένας Σουηδός συνάδελφος ο οποίος έχει πάρει πρωτοβουλίες, μία συνάδελφος, έχει πάρει πρωτοβουλίες για το θέμα των αναστολέων, έχει πάρει υποσχέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ευχαριστούμε, Κρίς Ντέιβις τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίσατε, Υπουργέ. Θα ήθελα να σχολιάσω δύο ζητήματα. Το πρώτο ε, σχετίζεται με την εφαρμογή του ενωσιακού περιβαλλοντικού προγράμματος ε, με όσους όρους για όλους και κυρίως για την ορθότητα της εφαρμογής. Ενομοθετούμε και ε, τελικά η εφαρμογή της νομοθεσίας ποικίλει από κράτος σε κράτος και ενδέχεται τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ε, ε, ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες να δυσκολεύονται το ώστε να φέρνουν σε πέρα με ικανοποιητικό τρόπο τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις παραδείγματος χάρη σε σχέση με άλλες χώρες. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Ε, αναρωτιέμαι εάν ε, υπάρχει όμως και έλλειψη συνοχής ε, ως προς την προσέγγιση των κρατών μελών. Η νομοθεσία μιλάει για αποτρεπτικές και ε, αναλογικές κυρώσεις. Υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο λιγμών, εκεί ήθελα να καταλήξω, για την εφαρμογή από πλευρά των κρατών μελών ε, και ήθελα να σας ρωτήσω πότε είναι η τελευταία φορά που συζητήθηκε αυτό το ζήτημα της ανομοιόμορφης εφαρμογής του, ε, της νομοθεσίας στο Συμβούλιο ή να το πω και πιο ομά γιατί δεν το θέτεται αυτό το ζήτημα. Δεύτερον, για το θέμα της πλαστικής ε, σακούλας. Ε, υπάρχει το ζήτημα των πλαστικών αποβλήτων ε, που τίθεται γενικότερα. Υπάρχουν ε, πολλοί από πλευράς βιομηχανίας που θα μας πούν ότι από πλευράς διοξιδίου του άνθρακα, παραδείγματος χάρη, Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές ε, άλλα εναλλακτικά είδη σακούλας ε, που επιφέρουν και μεγαλύτερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με τις πλαστικές σακούλες. Εγώ να ρωτιέμαι ποιο θα είναι το μέλλον της συζήτηση ε, για αυτό το ζήτημα στο Συμβούλιο. Ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρος, κυρία Σατοχάση. Ευχαριστώ τον Υπουργό που ήρθε σήμερα μαζί μας για να συζητήσουμε ένα τόσο ευρύ φάσμα ζητημάτων, όπως είδαμε στην εισαγωγική σας παρουσίαση. Αναφερθήκατε στο κλιματικό πακέτο που δημοσίευσε ε, χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκομίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πακέτο για τις κλιματικές αλλαγές ε, ως φιλόδοξη. Αναρωτιέμαι, ε, εντάξει δικό της είναι το πακέτο, δική της είναι η πρόταση, τι άλλο θα μπορούσαν να πούν. Όπως είπε η Λίντα Μακέβαν όμως, συμφωνώ και εγώ, είναι απογοητευτικό το αποτέλεσμα και δημοσιεύματα τύπου σήμερα αναφέρουν ότι Απογοητεύθηκαν και διπλωματές από τις τρίτες αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο ελπίζω να καταβάλει κάθε δυνατή ε, προσπάθεια ώστε να ενισχυθεί παραδείγματο χάρη η βαρύτητα της ενεργειακής αποδοτικότητας και η βαρύτητα των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών. Έχω δύο ερωτήσεις να σας θέσω ε, που σχετίζονται ε, με πιο ε, λεπτομερή νομοθετική ρύθμιση περιβαλλοντικών ζητημάτων. Πρώτον, ξέρουμε ότι ο τομέας όπου αυξάνονται πάρα πολύ γρήγορα οι εκπομπές είναι οι μεταφορές. Υπάρχουν πολύ σημαντικά νομοθετήματα που έχουν ήδη δρομολογηθεί ε, που στόχο έχουν να ε, αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των αυξανόμενων εκπομπών. Η νομοθεσία ILOC, ε, ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα, περί του οποίου δεν, υπάρχει, δεν έχει ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατάξει μία θέση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει την ιδέα να υπάρξει ένα ανώτατο όριο για τα καύσιμα που προέρχονται από βρόσιμες πρώτες ύλες. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επίσης αλλαγές στην έμεση χρήση γης και παράγοντες που σχετίζονται με ιδιαίτερα με τα καύσιμα ή με τις πρώτες ύλες. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τις προθέσεις της ελληνικής ε, προεδρίας. Θα εργαστείτε σκληρά ώστε να επιτύχετε κοινή θέση για το, ε, τον φάκελο, για το πακέτο ILOC. Δεύτερον, οδηγία για τα καύσιμα. Ε, άλλη μια απογοήτευση, πηγή απογοήτευση στο πακέτο που δημοσίευσε χθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάναμε εδώ μια ανταλλαγή απόψεων με του εκπροσώπους της Επιτροπής και μιλήσαμε για το εξή ζήτημα. Στο πακέτο κλιματικών αλλαγών προπενταετίας ε, η οδηγία για τα καύσιμα είναι η μόνη που δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Θέλω να γνωρίζω λοιπόν εάν η ελληνική προεδρία υποστηρίζει την εφαρμογή της οδηγίας ε, για τα καύσιμα και αν υποστηρίζει την λήψη ε, της ε, απαιτούμενης απόφασης. Τρίτον, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Εχθές άκουσα ότι αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας. Όμως ο, πράσινος, ο συνάδελφος από τους πράσινους Έλληνα συνάδελφος από τους Πρασίνους, ε, έκανε την ερώτηση στον Υπουργό Υγεωργίας και εκείνος είπε ότι όχι, είναι αρμοδιότητα ε, του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Λοιπόν, θα ήθελα πολύ να ξέρω ποιανού αρμοδιότητα είναι η γενετικά τροποποιημένη στην ελληνική κυβέρνηση. Ξέρετε, την περασμένη εβδομάδα με συντριπτική πλειοψηφία το Κοινοβούλιο καταψήφισε την έγκριση ενός ε, ε, μιας νέας ποικιλία αραβοσιτού 1507 της Pioneer γενετικά τροποποιημένης ποικιλία διότι ε, αυτό συνιστά υπέρβαση των εκτελεστικών ή εφαρμοστικών αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βάσει των πληροφοριών που έχω προτίθεται η Ελληνική Προεδρία να θέσει ως σημείο α στο επόμενο εκοφήν αυτό το ζήτημα. Θα ξέρουμε επίσης ότι εσχάτως ε, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε την ε, έγκριση της γενετικά τροποποιημένης ποικιλία ε, της πατάτας φλόρα διότι ενέχει παρεμφερή κίνδυνο, υποθέτω. Ποια είναι η άποψή σας και πώς θα επιτύχετε συμμόρφωση με την νομοθεσία για τους γενετικά τροποποιημένους. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ιάννα Ρόσμπαχ, ε, σύντομα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ που ήρθατε σήμερα εδώ. ιδιαίτερο για την ε, για το ευρύτατο πεδίο των θεμάτων που καλύψατε με την παρουσία σας, παρουσίασή σας και την ενέργεια ιδιαίτερο που με ενδιαφέρει. Εγώ είχα κοιτάξει τα θέματα αυτά εν συντομία. Παρατηρώ λοιπόν ότι η Ελλάδα καταναλώνει ενέργεια για την θέρμανση των ιδιωτικών κατοικιών ίση με αυτή της Φινλανδίας. Πράγμα το οποίο με οδηγεί σε σκέψεις. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι για να χρησιμοποιείτε λιγότερη, να καταναλώνετε λιγότερη ενέργεια στην Ελλάδα. Αλλά δεν ήρθαμε μόνο να μιλήσουμε γι' αυτό. Ε, πρέπει να συζητήσουμε και το γενικότερο θέμα της ε, ενεργειακής εξάρτησης και τον περιορισμό των, ε, της χρήσης των καυσίμων ορυκτής προέλευσης. Πρέπει δηλαδή να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση της αιωλικής ενέργειας. Γιατί υπάρχουν διάφορες μορφές τεχνολογίας που μπορούν να μας απασχολήσουν. Η πλαστική σακούλα δεν είναι μόνο απόβλητο. Μπορεί να είναι ενεργειακή πηγή. Άρα λοιπόν μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να επαναξιοποιούμε τα πράγματα αντί να τα πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων. Υπάρχουν τρόφιμα, ε, τροφές, ε, τα υπολείμματα των τροφών, αυτά που μένουν στο πιάτο μας, τα οποία μπορούμε επίσης να αξιοποιήσουμε σαν μια βιώσιμη μορφή ενέργειας. Μιλήσατε για την ατμοσφαιρική ρήπανση και γενικότερα τη ρήπανση. Νομίζω ότι η ρήπανση δεν αφορά μόνο την ε, ατμόσφαιρα. Ιδιαίτερο φαινόμενο ρήπανσης έχουμε από τον κλάδο της ναυτιλίας. Η Ελλάδα, μεγάλο ναυτικό κράτος, έχει και πολλά πλοία με ελληνική σημαία και ως εκ τούτου πιστεύουμε θα πρέπει να αναλάβει δράση για την προστασία της βιοπικιλότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος σε όλα αυτά τα θέματα ε, που αφορούν πάνω από όλα για σας την ε, Μεσόγειο. Θα ήθελα επίσης να συζητήσουμε, να μας πείτε αν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σχέδια, έργα που ενδεχομένως αναπτύσσονται σε συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών κρατών. Εγώ προέρχομαι από τη Δανία. Ξέρετε, ε, η γειτονική μας περιοχή είναι η Βαλτική, όπου όλα τα κράτη έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα όλοι οι κανόνες ε, που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύουν και στα κράτη. Αυτά δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα δηλαδή. Εσείς όμως που έχετε γείτονες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορείτε να βοηθήσετε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και την προστασία της βιοποικιλότητας της ε, Μεσογείου. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου και ευχαριστώ πολύ ιδιαίτερα για την έμφαση και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίσετε τη βιοποικιλότητα. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε τον Καρλ Χάιντς Φλόρενς ο οποίος έχει προσκαλέσει ε, συνεργάτες από την εταιρεία του η οποία ασχολείται ιδιαίτερως με την υγεία των ε, ζώων, για την οποία είναι και αρμόδια η Επιτροπή μας, εάν οι πληροφορίες μου είναι σωστές, αυτή είναι η δουλειά σας, ε, ασχολείστε ε, με θέματα υγείας των ζώων στην Αμερική αλλά και την Ευρώπη. Καλώς ήρθατε λοιπόν και εσείς. Συνεχίζουμε του συντονιστέ. Και παρακαλώ τον κύριο Αγκουράκη να λάβει το λόγο αν προφέρω σωστά το όνομά σα και, με ζητώ, και ζητώ συγγνώμη αν τυχόν είναι λάθος. Ε, όχι, όχι, μια, χαρά το μεταφράσατε, το προφέρατε, πολύ σωστά. Ε, η, η, εκτίμα, η εκτίμησή μας είναι ότι το πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας, τα μέτρα που καλείται ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της να εφαρμόσει στην τελευταία Προεδρία, άμα θέλετε, πριν ε, τις ε, ευρωεκλογέ σηματοδοτούν μια παραπέρα ε, επίθεση ε, τόσο στα εργασιακά και δημοκρατικά δικαιώματα και κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων όσο και όσον αφορά την κατάσταση ε, που επικρατεί στον τομέα του περιβάλλοντος. Το σημειώνουμε αυτό γιατί όπως αναφέρθηκε και εισαγωγικά από την Ελληνική Προεδρία το όλο πρόγραμμα βεβαίως και κινείται στα πλαίσια και της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και της ε, οικονομικής διακυβέρνησης και ε, του Συμφώνου για την σταθερότητα και της απασχόλησης, δηλαδή αυτών των πολύ σκληρών πολιτικών που έχουν ε, οδηγήσει σε μια ε, απερίγραπτη κατάσταση σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αναφέρουμε στα 27 εκατομμύρια ανέργους, αναφέρουμε στα 100 στους 100 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στα όρια της φτώχειας. Επίσης ε, θεωρούμε ότι στο όνομα της αντιμετώπισης των ε, περιβαλλοντικών προβλημάτων αλλά στην πραγματικότητα για να εξυπηρετηθούν ε, τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και αν θέλετε και σε μια προσπάθεια να βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την καπιταλιστική κρίση στην οποία βρίσκεται είχαμε την εφαρμογή των, της αρχής ορυπαίνων πληρώνει και, και τη δημοπρασία όσον αφορά τους ρήπους που αποδείχτηκε ότι στην ε, πραγματικότητα χρησιμοποιήθηκαν για την εκτόξευση των κερδών των ε, μεγάλων ε, μονοπωλιακών ομίλων και όχι για την βελτίωση των συνθήκων και κυρίως της γενικότερης κατάστασης των εργαζομένων. Και πραγματικά, επειδή δεν έγινε και καμία ιδιαίτερη αναφορά και επειδή συζητήθηκαν και γενικά διάφορα πράγματα, θα ήθελα να, να αναρωτηθώ, ας πούμε, τι μπορούν να πιστεύουν οι Έλληνες εργαζόμενοι ή οι εργαζόμενοι στην Ισπανία από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όταν ξέρουμε ότι στην Ισπανία έχει χάσει μια φούσκα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και είναι χιλιάδες αυτοί που έχουν χάσει τα λεφτά τους, στην Ελλάδα ακυρώνονται χιλιάδες άδειες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διότι λέει, δεν αποδίδουν πλέον και ταυτόχρονα όμως έχετε μια εκτείναξη των τελών ΑΠΕ στους λογαριασμού της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία εκτείναξη βεβαίως συμβάλλει και αυτή ώστε δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες και πιστεύω είναι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες στη Νότια Ευρώπη οι οποίες ε, στερούνται του βασικού δικαιώματος να έχουν πρόσβαση ε, στον ηλεκτρισμό, στην ηλεκτρική ε, ενέργεια. Εμείς θεωρούμε ότι η συνέχιση αυτής της πολιτικής θα, θα βλάψει ακόμα περισσότερο την γενική κατάσταση. Σημειώνουμε ότι παρά την εφαρμογή της Ευρώπης 2020 η ανεργία αυξάνει και τέλος δεν μπορώ να μην ε, αξιοποιήσω αυτή την, την ευκαιρία για να επισημάνω την απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει στο τομέα της επεξεργασίας ε, σκουπιδιών στην Ελλάδα. Είμαι μέλος της Επιτροπής ε, Αναφορών. Υπήρχε μια επίσκεψη το Σεπτέμβρη και η Επιτροπή είδε μια κατάσταση που, ξεκινάει, που υπάρχει σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Ιδιαίτερα θέλω να κάνω αναφορά στην κατάσταση που υπάρχει με μια πολύ μεγάλη χωματερή στην, στην Αθήνα ε, που ταλαιπωρεί για 50 χρόνια τους εργαζόμενους και δεν φαίνεται να υπάρχει καμία προοπτική να, λυθεί το πρόβλημα αυτό. Και τέλος να αναφερθώ σε μια παράδειγμα κατάσταση που υπάρχει στο Δήμο της ε, Ερμιώνης μιας και έγινε λόγος για την ε, θαλάσσια στρατηγική και για την μπλε ανάπτυξη. Εκεί με ευθύνε τη ελληνική κυβέρνηση υπάρχει μια μεγάλη πολυεθνική που κατασκευάζει ξενοδοχεία, ρηπαίνει το περιβάλλον, έχει πάρει τι άδειε και έχει μεγάλη ευθύνη η ελληνική κυβέρνηση ε, για το ότι παραβιάζονται βασικοί κανόνε και βασικέ αρχέ. 50.000 τόνοι σκουπιδιών είναι πεταγμένα από εδώ και από εκεί, απειλείται το περιβάλλον. Ε, γιατί όλα αυτά για να εξυπηρετηθούν ε, τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, θα ε, κάνουμε το εξή τώρα. Συνονιθήκαμε τον Υπουργό να ακούσουμε όλου του ε, συναδέλφου για να κάνουν τι ερωτήσει του και να απαντήσει μετά. Παρακαλώ όμω του συναδέλφου να περιοριστούν μόνο στο 1,5 λεπτό. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Για να σα ακούσουμε όμω όλου, για να απαντήσει σε όλου. Ο Υπουργό, παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ο Καρλ Χάιντ Φλόρεν. Ένα λεπτό και 30 δευτερά. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα πράγματα. Ε, αναφερθήκατε στο, στη μεταφορά αποβλήτων, shipment of waste. Είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει. Έχουμε δει πόσο αδύναμη είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμη έναντι των κρατών μελών, διότι απλώς δεν έχουν εφαρμόσει νομοθεσία παλιά. Είναι κρίμα και είναι ντροπή και γι' αυτό παρακαλώ να μεριμνήσετε ώστε οι κανόνες που από κοινού έχει συμβολή στο Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο το όντι να υλοποιούνται. Το ίδιο αφορά άλλωστε και τις ε, σακούλες. Το έχουμε συζητήσει. Εάν δεν φροντίσουμε στην Ευρώπη να διαχωρίζουμε τα απόβλητα, τα σκουπίδια και ε, έχουμε πολύ περιορισμένα ποσοστά μέχρι 60-80% στην ανακύκλωση, τότε βεβαίως θα έχουμε σοβαρά προβλήματα και με τις ε, σακούλες. Θα ήθελα επίσης να πω ότι είμαι βέβαιος ότι θα κάνετε το καλύτερο δυνατό στην ε, Προεδρία σας και σας παρακαλώ να παραμείνετε στο δυνατόν πιο άτεγκτοι στην ε, υπόθεση των θεμάτων. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπε η κυρία Χάση. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να ε, προσπαθούμε να τροποποιούμε νομοθεσία όταν δεν ξέρουμε που θα μας οδηγήσει. Καλό θα είναι λοιπόν για το iLook να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί, γιατί τότε θα καταλήξουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά προβλήματα και ίσως τελικά να μεταθέτουμε τα προβλήματα στην επόμενη Προεδρία. Ευχαριστώ κύριο Αρσένης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας, εδώ πέρα, με την πράσινη κάρτα. Ε, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας και ε, θέλω να ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο και αυτή η Επιτροπή θα είναι στο πλευρό σας για κάθε θετική πρωτοβουλία που θα πάρει η Προεδρία και θα τη στηρίξουμε ε, με όλη μας την καρδιά. Ε, πριν από κάποιο διάστημα ε, είχα καταθέσει μια ερώτηση ε, για την εφαρμογή, για την παραβίαση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών ε, οδηγιών αλλά και των διεθνών προδιαγραφών κατά τις σεισμικές έρευνες για πετρέλαιο στα, στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Είχατε πει τότε ότι το να ζητάω ε, κανόνες, την εφαρμογή των κανόνων, πα, ε, να βάζω την εφαρμογή των κανόνων πάνω από την εξόρυξη πετρελαίου με κάνει επικίνδυνο για τη χώρα. Ε, στην, ε, είναι γνωστό και σας αναγνωρίζετε ότι η βασική σας, βασική σας πολιτική ατζέντα είναι η, ακριβώς η προώθηση της εξόρυξης πετρελαίου ως βασικό στατικό, ως ε, προϋπόθεση για να έχει η χώρα ένα, ένα μέλλον, όπως πολύ συχνά λέτε. Και ήσασταν και γι' αυτό το λόγο, φαντάζομαι, και εναντίον του, του backloading στο ETS. Ήθελα να σας ρωτήσω, με δεδομένο αυτές τις θέσεις, πώς θα μπορέσετε να ηγηθείτε του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος, ε, στη προσπάθεια της Ευρώπης αυτή την κρίσιμη περίοδο να επεξαρτηθεί από το πετρέλαιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε κυρία Εστρέλα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Υπουργέ, καλώς Θα ήθελα να σε ευχηθώ κάθε επιτυχία για την Προεδρία. Τον Οκτώβρη στην Κορέα θα γίνει η συνέλευση των συμβαλωμένων μερών της Σύμβασης του ΟΗΕ για την βιοπικιλομορφία. Ε, είναι πολύ σημαντικές οι διαπραγματεύσεις διότι στόχος είναι να ενισχύσουμε την προστασία των οικοσύστηματων και διαφόρων ε, υποεξαφάνιση ειδών. Πέρυσι είχα την ευκαιρία να προεδρεύω της αποστολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παρακολουθούσε ε, την COP στην Ινδία, την συνέλευση των συμβαλωμένων μερών στην Ινδία και είδαμε ότι σημειώθηκε πολύ σημαντική πρόοδος ε, σε σχέση με τη χρηματοδότηση όλος ιδιαιτέρως. Ε, δηλαδή δεσμεύτηκαν τα συμβαλόμενα μέρη να διπλασιάσουν την προσπάθεια που κάνουν μέχρι το 2015 στις αναπτυσσόμενες χώρες λαμβάνοντας υπόψη το θέμα της ε, διάσκεψης που είναι η βιοπικιλομορφία για μια βιώσιμη ανάπτυξη και λαμβάνοντας υπόψη ε, επίσης ε, το πρόγραμμα της ελληνικής προεδρίας στο οποίο εμπίπτει και η προετοιμασία αυτής της σημαντικής διάσκεψης σας ερωτώ ποιες θα είναι οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις της παγκόσμιας αυτής διάσκεψης τον Οκτώβρη στην Κορέα στην Κορέα. Ευχαριστώ, ο κύριος Δανέλης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Θέλω να ευχηθώ στην Ελληνική Προεδρία να ασκήσει το ρόλο της προθετικά και αποτελεσματικά στην ε, πρόθεση και την επίλυση ζητημάτων που απασχολούν το κοινό μας σπίτι. Και βεβαίως πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σταθεί επικοδομητικά στο πλευρό σα στι προσπάθειε που θα καταβάλλετε. Θέλω να συγχαρώ την Ελληνική Προεδρία γιατί συμπεριέλαβε στι προτεραιότητέ τη την γαλάζια ανάπτυξη και συνολικά την θαλάσσια οικονομία. Ε, και ως ο εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο για την γαλάζια ανάπτυξη ε, θα ήθελα να σα ζητήσω, παρότι έχω αντιληφθεί ότι δεν θα είστε εσεί ο βασικό στον συντονισμό των θαλασσίων πολιτικών, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ένα ζήτημα όμως κλειδί για την πρόθεση της γαλάζιας ανάπτυξης είναι το, το εξή, που εσείς αντιλαμβάνεστε και εξαιτία του ρόλου σας, αλλά και των ευαισθησιών των προσωπικών που έχετε. Ε, όσο αυξάνονται οι, οι εντάσεις, όσο αυξάνονται οι χρήσεις ε, του θαλάσσιου ή του παράκτιου περιβάλλοντος, ε, τόσο δημιουργείται μεγαλύτερη ε, ε, ανάγκη ώστε να έχουμε μια συστηματική και συντονισμένη και βεβαίως σχεδιασμένη διαχείριση του θαλάσσιου και του παράκτιου περιβάλλοντος. Αυτό θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο και για την προστασία του, εξαιρετικά ευαίσθητου θαλασσίου περιβάλλοντος και για την διασφάλιση της βιωσιμότητας κάθε αναπτυξιακής διαδικασίας. Έτσι λοιπόν κλειδί σε αυτή την υπόθεση είναι ο θαλάσσιος σχεδιασμός. Όμως το επειδή έχουμε ήδη μπει στον πρώτο τρίλογο, ολοκληρώθηκε και πάμε στον δεύτερο τις επόμενες μέρες, η εικόνα που εισπράττουμε από το Συμβούλιο είναι απογοητευτική. Ε, η αντίληψη του Συμβουλίου είναι εξαιρετικά αρνητική στο να προχωρήσουμε σε ένα ουσιαστικό ε, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και γι' αυτό το λόγο το επισημαίνω σε εσά και θα ήθελα την εμπλοκή σας με όποια πρωτοβουλία θεωρήσετε ότι μπορείτε να έχετε θεσμικά και νομίζω ότι θα, θα βοηθήσει εξαιρετικά στην ποιοτική βελτίωση των προτάσεων του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε δεν είναι... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να πάρω το λόγο σχετικά με την αμφισβητούμενη εμπολής πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αδειοδότηση της καλλιέργειας του καλαμποκιού ΜΟ 1017. 1507 της Ντουιπό η πρόταση αυτή αντιπροσωπεύει για την ε, ελληνική προεδρία ένα γρίφο. Ένα γρίφο νομικό αλλά καταλαβαίνω και ένα γρίφο πολιτικό. Υπάρχει το θέμα του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας, δεν ξέρω πότε θα συζητηθεί το θέμα, δεν ξέρω αν θα συζητηθεί το θέμα. Πάντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απορρίψει με μεγάλη πλειοψηφία την ιδέα της αδειοδότησης αυτού του ε, γενετικά τροποποιημένου ε, οργανισμού γιατί θα προκαλέσει συνέπειες καταστροφικές σε ορισμένες πεταλούδες, σε ορισμένα είδη πεταλούδας. Λοιπόν, διαρωτώ με, ε, τι συσχετισμός δυνάμεως θα δημιουργηθεί στο εσωτερικό του Συμβουλίου ε, αν αδειοδοτήσετε, δεχθείτε αυτήν την μικρή εξαίρεση, τότε ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης γύρω από το θέμα των γενετικά τροποποιημένων γενικά. Ευχαριστώ. Ακούσαμε όλους τους εγγεγραμμένους για ερωτήσεις. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι εχθές ε, συζητήσαμε την πρόταση για τους στόχους 2030 με την παρουσίαση με μείωση των εκπομπών του διοξιδίου 27% συνολικό πόρο, συνολικούς πόρους από ανανεώσιμες πηγές που είναι μάλλον καταφληπτικός στόχος διότι δεν έχει τίποτα το συγκεκριμένο μέσα. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερο δυναμικό και για απασχόληση εάν κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις και μπορέσουμε να κάνουμε τη μετα... μετάβαση από τη βιομηχανία που χάνουμε στους νέους κλάδους ε, που μπορούν να δημιουργηθούν. Και πρέπει να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε με επενδύσεις σίγουρες που μπορούν να αναπτυχθούν. Παρακαλώ να λάβετε και αυτό υπόψη σαν παρατήρηση. Και στο επίκεντρο βέβαια των ε, αγώνων μας για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής είναι το σύστημα των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα, ξέρετε, ε, του ε, εκπομπών καυσαερίων, ξέρετε ότι αυτό είναι το καλύτερο μέσον που έχουμε σε θέσή μας, αλλά το άριστο μέσον θα ήταν βέβαια ο φόρος στο διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο όμως δεν είναι... Ε, δεν έχει γίνει δεκτό. Έχουμε λοιπόν τη δεύτερη καλύτερη λύση, το σύστημα των ανταλλαγών εκπομπών και νομίζω ότι κάποια πράγματα μπορεί να μας διδάξει το Ηνωμένο Βασίλειο με το Carbon Flow Price μια ιδέα καλή, η οποία όμως σημαίνει ταυτόχρονα και μια δικλίδα ασφαλείας προς τα πάνω, έτσι ώστε να μην ε, κινδυνεύουμε με σοβαρέ αντιπαραθέσει μεταξύ Βουλίου και Κοινοβουλίου που δεν θα οδηγούν σε αποτέλεσμα, αλλά να υπάρχει δυνατότητα της προσαρμογής της τιμή. Όταν δηλαδή ε, δεν έχουμε αρκετά αποτελέσματα από τι ανταλλαγέ, να προσαρμόζονται οι τιμέ του πετρελαίου, του φυσικού αερίου ε, και αναλόγως να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τις τιμές εκείνων των ενεργειακών πόρων οι οποίοι δεν μας κοστίζουν σε εκπομπές. Αυτό για να προσθέσουμε και τις θέσεις εργασίας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν μπορεί να συνεχιστεί η εφαρμογή του συστήματος των ανταλλαγών. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα σοβαρό προγραμματισμό και σχεδιασμό για να κερδίσουμε και την βιομηχανία, το γενικά τον κλάδο που εφαρμόζει τις, ε, τα συστήματα αυτά και Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε μία μέση τιμή για τα πιστοποιητικά διοξιδίου του άνθρακα μέχρι τον Απρίλιο. Αυτή είναι η δική μου προσωπική τοποθέτηση. Δεν σας ζηλεύω, δεν σας φθονώ για το έργο που προλαμβάνετε να διαπραγματευτείτε τους στόχους 2030 για, ε, με το Συμβούλιο. Πρέπει ωστόσο να συμπληρώσω στι παρατηρήσει αυτέ ότι η Επιτροπή, και ιδιαίτερα ο πρόεδρο Μπαρόσο, έχουν αγνοήσει τι θέσει του Κοινοβουλίου. Έχουν περάσει μήνε όπου τα θέματα αυτά κυκλοφορούν μεταξύ Επιτροπή Περιβάλλοντο και Επιτροπή Βιομηχανία, των δύο άκρων δηλαδή, και, μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια, και μπορέσαμε να οδηγηθούμε σε μια απόφαση που έλεγε 40% μείωση του εξιδίου του άνθρακα, 40% αποτελεσματικότητα στην ε, αξιοποίηση τη ενέργεια που θα συμπλήρωνε το πρόγραμμα και το θα το καθεστούσε και ένα πρόγραμμα παραγωγή θέσεων εργασία για τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, για να εξασφαλιστούν περισσότερε θέσει εργασία, για να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση του ενεργειακού μα κλάδου. Και όπω είπαμε, ανανεώσιμε πηγέ, αλλά οι στόχοι πρέπει να είναι όχι μόνο ευρωπαϊκοί και εθνικοί. Αλλιώ τίποτε δεν μπορεί να χρησιμεύσει. Γι' αυτό λοιπόν φαντάζομαι ότι θα έχετε σκληρή δουλειά στο Συμβούλιο των Υπουργών περιβάλλοντος. Αυτά που είδαμε χθες από την Επιτροπή μπορεί σαν προθέσεις να ακούγονται ωραία, αλλά ήταν πολύ ασαφή. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τι τελευταίε παρατηρήσει του κυρίου Προέδρου, ο οποίο προσπάθησε και να συμπυκνώσει τον προβληματισμό που υπάρχει. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι από τη θέση της προεδρεύουσας χώρας θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει το θεσμικό <coughs> πλαίσιο, ώστε να προωθήσουμε ως το δυνατόν πιο φιλόδοξες περιβαλλοντικές θέσεις της Ένωσης σε όλα τα ζητήματα. Και σας μιλώ εκ μέρους του συνόλου των Ελλήνων Υπουργών. Διότι αυτή είναι μια κατεύθυνση προς την οποία θέλουμε να βαθίσουμε αντιλαμβανόμενοι απολύτως ότι το μέλλον της Ένωσης δεν μπορεί παρά να στηριχθεί στη συμβίωση της αηφορίας, της βιωσιμότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε δράσεις πράσινης ή γαλάζιας ε, κατεύθυνσης και ταυτόχρονα στην διατήρηση, και νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, της ανταγωνιστικότητας και της βιομηχανίας, αλλά επιτρέψτε μου να πω και κάτι που συνήθως το αγνώμαι την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν τον εργοδότη σχεδόν του 90 με 95% των Ευρωπαίων εργαζομένων. Θέλω λοιπόν να σημειώσω πως ε, προσδοκούμε ως Προεδρία και εγώ ως Προεδρεύων του Συμβουλίου Περιβάλλοντος τη στήριξη των Ευρωβουλευτών των αντίστοιχων επιτροπών και ιδιαίτερα της πολύ σημαίνουσας Επιτροπής Περιβάλλοντος, διότι θεωρώ πως οι στόχοι μας είναι κοινοί και ενιαίοι. Και επιτρέψτε μου, όχι πια ως Προεδρία, αλλά ως χώρα να σημειώσω, ότι νομίζω πως από την παγκόσμια νομισματική κρίση και ιδιαίτερα από την κρίση που έχει χτυπήσει την Ευρώπη και ειδικά τις χώρες του Νότου, ελπίζω όλοι να έχουν βγάλει τα συμπεράσματα του πώς πρέπει να αποφεύγουμε φούσκες και πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση όλων αυτών των παραμέτρων με σοφροσύνη και με προοπτικές μέλλοντος. Επιτρέψτε μου λοιπόν κύριε Πρόεδρε να ξεκινήσω από εσά κάνοντας μια τέτοια συνολική τοποθέτηση. Για τον κύριο Λίζε, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την ε, επανάληψη της αλληλεγγύης προς τον ελληνικό λαό, πρέπει να σας πω ότι θεωρούμε πως βρισκόμαστε ήδη στο τέλος του δύσκολου δρόμου και δικαιούται πια ο Έλληνας πολίτης να διεκδικεί την θετική ανταπόκριση στις θυσίες τις οποίες έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια. Και χαιρόμαστε πράγματι γιατί οι εκπρόσωποι των λαών της Ευρώπης, οι ευρωβουλευτές, έχουν σταθεί δίπλα μας. Θέλω να σημειώσω ότι το ζήτημα της συναπόφασης, του governance, είναι πραγματικά ένα μεγάλο θέμα. Θεωρούμε πως θα πρέπει με γνώση την εμπειρία που αποκτήσαμε στο παρελθόν να συνειδητοποιήσουμε ότι αν θέλουμε η Ευρώπη να αποκτήσει αυτό που φιλοδοξούσε και συνεχίζει να φιλοδοξεί, δηλαδή να αποτελέσει ηγέτιδα δύναμη, τόσο στα ζητήματα της οικονομικής αποτελεσματικότητας, όσο και στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος τότε η μόνη διέξοδος είναι ο ένας να ακούει τον άλλον. Και αναφέρομαι στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Διότι στο τέλος της ημέρας αυτός που υφίσταται τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα είναι ο Ευρωπαίος πολίτης, ο οποίος πολλές φορές ορθά αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τον τρόπο που λειτουργούμε. Θεωρώ λοιπόν ότι εν και των επερχόμενων ευρωεκλογών έχουμε χρέος όλοι μας να δώσουμε αυτό το νέο μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι εδώ, είναι παρούσα, είναι η μόνη διέξοδος για τους λαούς, είναι η μόνη διέξοδος για να συνεχίσουμε να έχουμε μια ηγέτιδα δύναμη στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και θα πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση να δουλέψουμε όλοι μας. Η κυρία Μακαβάν ε, ε, ε έβαλε το ζήτημα του κατά πόσον η Προεδρία θα στηρίξει βελτιώσεις στην πρόταση της, ε, ε της Επιτροπής για το ε, Κλιματική Αλλαγή Ενέργεια 2030. Πρέπει να σας πω ότι η Προεδρία, καλός ή κακός, έχει το συγκεκριμένο ρόλο που έχουν όλες οι Προεδρίες. Στόχος της είναι να συντονίζει, να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων και ουσιαστικά να λαμβάνει υπόψη της τις θέσεις όλων των κρατών μελών. Κατά συνέπεια πρέπει να σας πω ότι εμείς θα επιδιώξουμε να βρούμε συνενέσεις που θα στοχεύουν, επαναλαμβάνω, στον ταυτόχρονο, στην ταυτόχρονη ελοπίση και των δύο στόχων. Προστασία από κλιματική αλλαγή και διατήρηση της ε, ε, ε, ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας σε επίπεδο μεγάλων επιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιτρέψτε μου εδώ να τονίσω κάτι που συνιστά προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας και που το αναφέραμε κατά την παρουσίαση την χθεσινή ε, στην Επιτροπή Ενέργειας. Το ζήτημα της προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών, των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος, όταν έχεις απέναντί σου περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών που κινδυνεύουν από ενεργειακή φτώχεια, συνιστά επίσης μια πολύ μεγάλη πρόκληση στην οποία πρέπει να απαντήσουμε θετικά. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να τα βάλουμε στην φιλοδοξία μας να βελτιώσουμε θετικά τις προτάσεις που έχουν κατευθεί. Αναφορικά τώρα με τους ενδοκρινείς διαταράκτες, που είναι ένα εξειδικευμένο θέμα, ε, ε, ε, θέλω να, να σημειώσω ότι ασφαλώς αποτελούν ε, ε, ε, ουσίες εξαιρετικά υψηλής ανησυχίας με τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ωστόσο από όσο γνωρίζουμε δεν έχει ακόμη υποβληθεί σχετική πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τον κύριο Ντέιβις, το ζήτημα των επιθεωρήσεων. Πραγματικά το ζήτημα των επιθεωρήσεων γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι ένα θέμα που συζητείται πάντα όταν συζητούνται εφαρμοστικοί κανόνες σε όλους τους κανόνες εφαρμόζονται, αλλά ε, ε, εναπόκειται πια στην λειτουργία των κρατών μελών να έχουν τις συγκεκριμένες θετικές ή λιγότερο θετικές ε, αντιδράσεις. Πάντως από την πλευρά της δική μας θεωρούμε ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο όταν υιοθετούμε μια οδηγία ή έναν κανονισμό να έχουμε διασφαλίσει ότι η εφαρμογή του θα είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης. για τις πλαστικές σακούλες πραγματικά θεωρώ πως έχει μεγάλη σημασία ε, ε, να το αντιμετωπίσουμε με την σοβαρότητα που ταιριάζει κυρίως σε σχέση ε, με την ρήπανση που προκαλεί στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η κυρία Χάση έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά σε κάτι που δεν το συζητήσαμε σήμερα και που επίσης θεωρούμε ως Προεδρείο ότι αποτελεί μεγάλη σπουδαιότητα ζήτημα τόσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και για τα ε, νοικοκυριά της οικογένειας μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος όλης της Ένωσης. Αναφερόμαστε στο ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής θωράκισης και κατοικιών και δημοσίων κτηρίων και επαγγελματικών κτηρίων. Πρέπει να σας πω ότι για μας αυτό ως Προεδρία συνιστά μία από τις τρεις-τέσσερις μέγιστες προτεραιότητες με την ταυτόχρονη ιδιότητα και του Υπουργού ε, ε, Ενέργειας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Σε εθνικό επίπεδο μάλιστα, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο προφανώς ότι πρέπει να κάνει ο καθένας περιγραφή της εθνικής του θέσης, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες να το πω, έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας που ξεπερνά τα 1,2 δις ευρώ. Είναι πρόγραμμα που τρέχει ήδη, που υλοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας σε πρώτη κατοικία και σε δημόσια κτίρια και φιλοδοξούμε στη νέα προγραμματική περίοδο να αυξήσουμε κατά τουλάχιστον 50% τα διαθέσιμα αυτά κονδύλια. Άρα το ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας πράγματι είναι μια σπουδαία προτεραιότητα. Για την ILUC πρέπει να σας πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ το, το, και το τελευταίο Συμβούλιο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ε, ε, εμείς θα διερευνήσουμε και θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνει η ιδιότητα της Προεδρίας ώστε να δούμε αν μπορούμε να έχουμε κοινή θέση αποδεκτή ε, από όλα τα κράτη-μέλη. για, τους, ε, για την οδηγία για τα καύσιμα. Πρέπει να σημειώσω πως ε, ε, στο χρονικό αυτό διάστημα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, εκπονείται μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναμένουμε τη σχετική μελέτη και τις επιπτώσεις και ε, εάν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας έχουμε τη δυνατότητα να το φέρουμε για συζήτηση, θα είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε για μια πολύ ουσιαστική συζήτηση στο Συμβούλιο και να προωθήσουμε το συγκεκριμένο ε, θέμα. Για το ζήτημα των γενετικά τροποποιημένων ε, οργανισμών. Τα θέματα της έγκρισης καλλιέργειας ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου των Υπουργών Γεωργίας και έχουν συζητηθεί στις αντίστοιχες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Θέλω όμως να επισημάνω τα εξής δύο σημεία. Πρώτον, προφανώς το Συμβούλιο είναι ενιαίο, ανεξάρτητα από τη σύνθεση υπό την οποία συζητείται κάθε συγκεκριμένο θέμα. Για την έγκριση της καλλιέργειας του γενετικά τροποποιημένου του, το Συμβούλιο οφείλει να εκφράσει τη γνώμη του ως προς την πρόταση της Επιτροπής ω 12 Φεβρουαρίου 2014. Και είμαι βέβαιος ότι θα το πράξει. Η δεύτερη παρατήρηση σχετίζεται με τη θέση της χώρας μου όσον αφορά την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και οφείλω να σας πω ότι συνεχίζει και θα συνεχίσει να είναι εξαιρετικά αρνητική προς αυτή την κατεύθυνση. Το ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας το έθεσε και η κυρία Ρόσμπαχ και ε, έχετε, έχετε δίκιο. Η Ελλάδα καταναλώνει όσο και η Φιλανδία. Είναι η ενεργειακά πιο σπάταλη χώρα της Ευρώπης. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει με αρκετές χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση σε άλλες χώρες. Άρα έχουμε κάθε υποχρέωση όλοι, ως εκπρόσωποι των λαών που μας εκλέγουν, να λάβουμε μέτρα ενίσχυσης της ε, εξοικονόμησης ενέργειας. Επιτρέψτε μου επίσης να φέρω σε γνώση σας το γεγονός ότι για παράδειγμα η ολική ενέργεια που αποτελεί μια σπουδαία καθαρή πηγή ενέργειας για την Ελλάδα έχει και θα συνεχίσει να έχει σημαντικές προοπτικές στην ε, χώρα μου, ιδιαίτερα στον νησιωτικό χώρο και όχι μόνο. Μάλιστα κατά σύμπτωση τον προηγούμενο μήνα είχα την χαρά ως Υπουργό Περιβάλλοντος να εγκρίνω τις περιβαλλοντικές μελέτες για περίπου 16 μεγάλα αιωλικά πάρκα περίπου χιλίων μεγαβάτ. Άρα αυτό δείχνει ότι έχουμε μπροστά μας και προσέλκυση επενδύσεων και πολιτική βούληση να προχωρήσουμε αλλά και ενδιαφέρον να υλοποιηθούμε συγκεκριμένες δράσεις. Για τις εκπομπές της ναυτιλίας ε, τοποθετήθηκα και είπα ότι είναι ένα σύνθετο θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε ε, η Προεδρία θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να, να, προχωρήσουμε ε, στα ζητήματα αυτά. Και ασφαλώς έχει μεγάλη σημασία να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα από τις γειτονικέ χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και νομίζω ότι η στενή συνεργασία που υπάρχει με όλες τις γείτονες χώρες, όχι μόνο ως Προεδρία, αλλά και ως Ένωση, θα μας βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Ε, για το ζήτημα της, ε, των προσβάσεων στον ηλεκτρισμό και λοιπό, ο κύριος Αγκουράκης έθεσε αρκετά θέματα. Αυτά έχουν απασχολήσει πάρα πολλές φορές το Εθνικό Κοινοβούλιο στην Ελλάδα. Δεν θα ήθελα να καταχραστώ το χρόνο σας για να κάνω ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα που έτσι καλώς συζητούνται στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Οφείλω όμως να σημειώσω ότι πραγματικά το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας είναι ένα σπουδαίο θέμα. Εδώ όμως να σας πω πως ε, στην Ελλάδα εδώ και τρία περίπου χρόνια εφαρμόσουμε μια κοινωνικά ευαίσθητη πολιτική στα ζητήματα της προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών, σήμερα στην Ελλάδα, σήμερα, το 15 με 20% του πληθυσμού χαμηλού εισοδήματος έχει ηλεκτρικό ρεύμα πολύ φτηνότερο από, το άλλο, από τα άλλα μέσα νοικοκυριά. Έχουμε δώσει μέσω του ονομαζόμενου κοινωνικού οικιακού τιμολογίου έκπτωση έως και 40% σε εξειδικευμένες κοινωνικές ομάδες. Μακροχρόνια ανέργους, άτομα με αναπηρία, τρίτεκνους, ανθρώπους που έχουν χαμηλό εισόδημα. Άρα σε αυτή την προσπάθεια ασφαλώς και πρέπει να προχωρήσουμε, όμως ήδη τα πρώτα βήματα έχουν γίνει. Θα μου επιτρέψετε επίσης να σχολιάσω το ζήτημα ε, των απορριμμάτων. Επίσης είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει το Εθνικό Κοινοβούλιο και πάντα απασχολεί και την Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Θέλω να διευκρινίσω τούτο. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ε, βρίσκεται σε μια ε, ε, όχι καλή θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και μάλιστα έχουν υπάρξει και συγκεκριμένες καταδίκες από το δικαστήριο. Να σας δώσω απλώς έναν αριθμό. Το 2005 είχαμε στη χώρα μου 1.125 χώρους που δεν ελέγχαμε ε, πώς πηγαίνουν τα απορρίμματα. Σήμερα οι χώροι αυτοί έχουν μειωθεί σημαντικά. Ε, έχουμε μόνο 78 ενεργούς χώρους ανεξάλλεκτης διάθεσης απορριμμάτων, οι λεγόμενες χωματερές, από τους οποίους χώρους αυτούς το 40% είναι σε πολύ μικρά νησιά, νησιά των 100, 200, 300 κατοίκων, για τα οποία θα πρέπει να δει κανείς πώς το αντιμετωπίζει εξειδικευμένα. Πάντως, για να μην μακρηγορήσω το συγκεκριμένο θέμα, να σας πω ότι όλες αυτές οι δράσεις είναι ενταγμένες σε χρηματοδοτικά σχήματα. Προχωρούμε όσο μπορούμε πιο σύντομα και όταν υπάρχει η αντίστοιχη βούληση από όλες τις πλευρές, τότε τα προβλήματα προχωρούν με την χρηματοδότηση και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Για το ζήτημα ο κύριος Φλόρενς της μεταφοράς απορριμμάτων των σακούλων ε, σακούλες, ανακύκλωση και i-look. Αντιλαμβάνουμε απολύτως τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορούν να υπάρχουν. Ε, οφείλω να σημειώσω πάντως πως η Προεδρία θα επιδιώξει συνενέσεις ε, σε όλα τα κράτη-μέλη έτσι ώστε όλα αυτά τα ζητήματα ε, να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ο κύριος Αρσένης έχει, έχει θέσει διάφορα θέματα. Να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Η Ελλάδα, όπως και κάθε χώρα, επιδιώκει να αξιοποιήσει το σύνολο των ενεργειακών της κοιτασμάτων. Αναφέρομαι στον ήλιο, τον αέρα, τη γεωθερμία, ε, τους υδρογονάνθρακες. Δεν θα αφήσουμε αναξιοποιητό κανένα ε, πλούτο ενεργειακό που μας έχει χαρίσει η φύση, επειδή ακριβώς κανένα κράτος σύγχρονα και αναπτυγμένο δεν αφήνει αναξιοποιητό τον πλούτο αυτό. Και βεβαίως οφείλω να υπενθυμίσω σε όλους μας την μεγάλη εξάρτηση της Ένωσης συνολικά ως οντότητας, ως συνολικής διεθνικής οντότητας, από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων απ' έξω. Από χώρες, από τρίτες χώρες. Τεράστια κονδύλια. Και θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρχει αντίρρηση αντί να κάνει εισαγωγή απ' έξω από τρίτες χώρες και να είσαι και ενεργειακά εξαρτημένος να επιδιώκεις, να αξιοποιείς τα ενδογενή ε, κοιτάσματα που έχει σε κάθε χώρα και αυτό πράττουν όλες οι χώρες. Υπάρχει μια βασική προϋπόθεση. Να εφαρμόζεις τις αυστηρότερες δυνατές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Και εδώ οφείλω να σας πω ότι η χώρα μου έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει απόλυτα και πιστά το σύνολο των ευρωπαϊκών προδιαγραφών που έχουν υπάρξει. Σε όλες τις δράσεις αξιοποίησης των κοιτασμάτων. Ε, των ενεργειακών ε, κοιτασμάτων κάθε είδους. κυρία Εστρέλα, για τα θέματα της βιοποικιλότητας της Κορέας ε, πραγματικά είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διεκδικήσει την πρωτοπορία στην προστασία της βιοποικιλότητας διότι ακόμη και για τους στιγνούς οικονομολόγους ακόμη και για αυτούς που μετράνε την ανθρώπινη ζωή ή την ύπαρξη του πλανήτη με ψυχρούς αριθμούς, ακόμη και στο επίπεδο το δικό τους, εάν μιλήσει κανείς, βλέπει ότι θα πρέπει και αυτοί να αλλάξουν εικόνα. Διότι η προστασία της βιοπικιλότητας αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο οικονομικό παράγοντα που φέρνει ευημερία σε λαούς και δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας. Ο κύριος Δανέλης αναφέρθηκε και χαίρομαι γι' αυτό, διότι αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μιας χώρας που γέννησε τον θαλάσσιο πολιτισμό όπως είναι η Ελλάδα. Βρισκόμαστε σε μία από τις πιο ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές του πλανήτη που είναι η Μεσόγειος θάλασσα. Και θεωρώ πως είναι μια καλή ευκαιρία η ελληνική προεδρία μαζί με την επερχόμενη την επόμενη Ιταλική Προεδρία να αναδείξουν σε μια σφιχτή, αποτελεσματική, οραματική, στρατηγική για τη γαλάζια ανάπτυξη το θέμα της αξιοποίησης του θαλάσσου περιβάλλοντος, περιβάλλοντος με όλες τις επιμέρους διαστάσεις του. Αλληλεία, τουρισμός, ναυτιλία, ενεργειακή πόρη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποκυματική ενέργεια μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Διαχείριση του παράκτου περιβάλλοντος. Πράγματι είναι μια σπουδαία δράση στην οποία όλες οι χώρες που έχουν ακτές πρέπει να δουν πώς θα υπάρξει συμβίωση του ευαίσθητου θαλάσσιου περιβάλλοντος με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που πάρα πολλές φορές επιβαρύνουν ε, το, το, το θαλάσσιο περιβάλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια καλή ευκαιρία με την Ελληνική Προεδρία και την ε, Ιταλική Προεδρία να διαμορφώσουμε άξονες στρατηγικής για ένα εξαιρετικά αναβαθμισμένο παράκτιο περιβάλλον για το καλό των Ευρωπαίων πολιτών η κυρία Οκονή, αναφορικά με το καλαμπόκι, ναι νομίζω ότι απάντησα. Είμαστε σε μια διαδικασία ε, ε, ε, αντιμετώπισης του θέματος με τον τρόπο που προανέφερα. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω σημειώσει άλλες παρατηρήσεις. Ε, φιλοδόξα να απαντήσω προσωποποιημένα σε όλες. Ελπίζω να το κατάφερα. Ε, εάν μου επιτρέπετε μόνο να κλείσω, θα ήθελα να πω πως επειδή πράγματι βρισκόμαστε σε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους της Ευρωπαϊκής Υπήρου και οι επερχόμενες ευρωεκλογές δεν είναι απλώς εκλογές για να εκλέξουν οι λαοί κάποιους ανθρώπους που θα τους εκπροσωπήσουν στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο στίχημα για το αν θα καταφέρουμε το πείραμα της Ευρώπης να το αντιμετωπίσουμε θετικά και να ξεπεράσουμε την κρίση που υπάρχει σε πάρα πολλούς τομείς. Πιστεύω βαθιά ότι τα ζητήματα της αηφορίας, της βιωσιμότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της αποτροπής των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μπορούν να βρουν τα καλύτερα μυαλά, τα πιο ανοιχτά αυτιά, τα πιο ανοιχτά μάτια στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στο Ευρωκοινοβούλιο. Γι' αυτό θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω θερμά για το ρόλο που έχουν, έχει παίξει ο κάθε Ευρωβουλευτής της Επιτροπής αυτής χωριστά, όλη η Επιτροπή και να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου και η επόμενη σύνθεση να είναι εξίσου θετική και εξίσου καλή. Εμείς ως Προεδρία ευελπιστούμε ότι θα δουλέψουμε μαζί χέρι-χέρι έτσι ώστε στο σύντομο χρονικό διάστημα να αντιμετωπίσουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ε, ήταν, πολύ όμορφα τα λόγια σας ως κατάληξη στην ομιλία σας, στον ευρωπαϊκό δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε, γιατί η Ευρώπη δεν είναι το πρόβλημα στην κρίση, αλλά η λύση στο πρόβλημα. Αυτό πρέπει πάντα να το υπογραμμίσουμε ότι η Ευρώπη είναι η λύση. Κανένα κράτος μόνο του δεν μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματά του. Όλα μαζί σε συνεργασία. Εσείς ιδιαίτερα δώσατε έμφαση στο ζήτημα της ενέργειας και είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτό. Αν από κοινού αναπτύξουμε διεθνικά προγράμματα και όχι μόνο μέσα στην Ευρώπη αλλά και αν στραφούμε προς τα έξω, Μεσόγειος Φερρυπίν, είναι λύσεις εκεί πάρα πολύ σημαντικές. Εύχομαι κάθε καλό στη χώρα σας. Έχετε δει με πολύ μεγάλες προκλήσεις αναλάβει να αντιμετωπίσετε. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Από τη δική μου την πατρίδα πάλι πρέπει να πω ότι ορισμένες εκφράσεις που έχω ακούσει και τοποθετήσεις με έχουν ε, κάνει να αισθανθώ όνειδος και ντροπή. Δεν μπορώ να στήσω συγγνώμη εκ μέρους γιατί δεν τις συμμερίζομαι, δεν τις έχω εκφράσει εγώ αυτές τις θέσεις, αλλά πρέπει να πω ότι με ντρόπιασαν. Η Ελλάδα είναι μια πολύ όμορφη χώρα. Δεν την έχω επισκεφθεί μόνο ως τουρίστας για τις για τις ε, διακοπές μου. Ε, ξέρω ότι έχει μεγάλο πολιτισμό και το μόνο μπορώ να πω κλείνοντας είναι ότι η Επιτροπή μας θα είναι στο πλευρό σας, θα σας υποστηρίζει. Ίσως και να σας σωθεί λίγο για να προχωρήσετε περισσότερο, πιο γρήγορα. Χαιρόμαστε πολύ για τη συζήτηση σήμερα. Θα είναι ενδιαφέροντες οι καιροί και σας εύχομαι κάθε επιτυχία και τύχη. Κάθε καλό λοιπόν και πάντα σας περιμένουμε κύριε Υπουργέ, κύριε Μανιάτη. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση σήμερα.